ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Θα προεδρεύσω στην αρχή γιατί ο πρόεδρος μας ε, έχει καθυστερήσει ε, η πτήση του. Είδατε την ημερήσια διάταξη, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Τώρα γιατί η διερμηνία υπάρχουν όλες οι γλώσσες εκτός από τη βουλγαρική και την κροατική και θα δώσω λίγα δευτερόλεπτα στους συναδέλφους διευμηνείς για το μήνυμά τους. Η... Η ελληνική Βρισκόμαστε στην 37η μέρα των κινητοποιήσεών μα λόγω τη επιβολή μονομερό ε, από τον Γενικό Γραμματέα Συνθηκών Εργασία στου Διερμηνεί και δεν θα χορηγήσουμε καμία υπέρβαση ωραρίου λόγω αυτή τη κινητοποίηση. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ε, au passage, quand même, avant d'entrer dans l'ordre du jour, Λοιπόν, πριν, ε, προχωρήσω να συγχαρώ τους Γάλλους, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει λυπάμαι για αυτό που έγινε χτες, αλλά θα τους υποστηρίξω στον τελικό. Τελικά στο ποδόσφαιρο είναι καλό ότι η Ευρωπαϊκή θα είναι η ομάδα που θα κερδίσει. Τώρα για την υπόλοιπη ημερήσια διάταξη έχουμε την έγκριση των πρακτικών της 7ης Ιουνίου, της 26ης και 25ης Απριλίου και της 21ης Ιουνίου. 28ης Ιουνίου σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξη. Υπάρχει ο τριγωνικός διάλογος για την εξωτερική υπηρεσία ασφάλειας και υγείας στην εργασία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Έγινε λοιπόν ένας τριμερής διάλογος στις 10 Ιουλίου Ε, με την Αυστριακή Προεδρία. Από ό,τι φαίνεται οι συζητήσεις έγιναν σε επικοδομητικό πνεύμα. Υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις σε μία σειρά πραγμάτων. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία και κομβικά τα οποία ακόμα μένει να αντιμετωπιστούν. Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται στις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου. Αυτά για τον τριγωνικό διάλογο. Περνάμε αμέσως τώρα στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, το θέμα το σχετικό με την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες ή σε μεταλλαξιογόνες ουσίες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει. Βρισκόμαστε στην τρίτη φάση, αν θέλετε, για τα προϊόντα αυτά και θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτριά μας, ε, την κυρία Τζέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπερήφανη που είμαι η του τρίτου τμήματος της οδηγίας αυτής για την προστασία των εργαζομένων ε, για τους κινδύνους ε, από την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Μέχρι τώρα νομίζω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά στα πλαίσια των δύο προηγούμενων ε, εξετάσεων του θέματος ορίσαμε 20 ανώτατα όρια για πάρα πολλές ουσίες και για 20 ουσίες, συγγνώμη, και τώρα για άλλες 5 στην τρίτη φάση για να εγγυηθούμε την προστασία των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνουμε σε επίπεδο κόστους με υπερβολικό τρόπο τις μικρομεσαίες. Νομίζω ότι μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά, επιτρέποντας με οργανωτικό και τεχνικό τρόπο να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Για το Βερίλιο, σαν παράδειγμα, προτείνεται επταετής περίοδος και όχι πέντε όπως η Επιτροπή προτείνει, χωρίς να αλλάξουμε όμως την, το ανώτατο ανεκτό όριο. Για να δώσουμε χρόνο προσαρμογής και να μην αναγκαστούν να πάνε σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα οι χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν προληπτικούς έκτακτους ελέγχους για την προστασία από τον περίλιο. Για το κάδμιο αφήσαμε το ανώτατο όριο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εκεί όπου είναι οι εγκαταστάσεις και υπάρχει έκθεση στο κάδμιο για επαγγελματικούς λόγους, είναι καρκινογόνο φυσικά το κάδμιο, τότε ο ιατρός ή η αρμόδια επί της υγείας αρχής θα παρακολουθούν συστηματικά και τεκμηριωμένα τους, ε, τους ανώτατους δείκτες καδμίου στα ούρα, δύο ε, μικρόγραμμάρια ε, και να φτάσουμε στο 0,004 μικρογράμμα στο μέλλον. Για το αρσενικό οξύ, τη φορμαλδεΐδη και το μόκα ή μεθυλένιο αλφα μικρό στην ουσία αφήνουμε τις, ε, τα όρια τα οποία έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα, για τις, ε, ανάλογα με τις επαγγελματικές κατηγορίες υπάρχει και σύμφωνη άποψη από πλευράς τους. Ε, υπάρχει μια ανάκαμψη οικονομική εδώ και αρκετό καιρό και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις που προσαρμόζονται στην οδηγία με κάποια κίνητρα σχετικά με το μέγεθος των επενδύσεών τους. Και τέλος, και εδώ υπάρχει θα θέλετε και μια ανάληψη υποχρέωσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να προχωρήσουμε ε, περιλαμβάνοντας ε, τα ε, κοιτοτοξικά φάρμακα, ιδιαίτερα στο πρώτο προσάρτημα, στο οποίο αν γίνεται αναφορά σε εργασίες οι οποίες οδηγούν σε έκθεση σε καρκινογόνες οξύς. Πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα που δουλεύουν στον τομέα της υγείας εκτίθενται σε επικίνδυνα φάρμακα, πολλές φορές α, ε, ε, α, μεταλλαξιογόνα, καρκινογόνα κτλ. Επίσης ε, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που χειρίζονται αυτά τα φάρμακα που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν λευχαιμία ή κάποιους όγους και οι νοσοκόμοι, οι, οποίοι, οι νοσοκόμες οι οποίες ε, ε, μεταχειρίζονται τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν διπλές ε, πιθανότητες διακοπής κοίησης. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επίσης εργαζόμενοι οι οποίοι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτοί και η οικογένειά τους και τα παιδιά τους ε, με αυξημένες παρουσίες όγκων, όπως επίσης και με αυξημένα ποσοστά διακοπής κοίησης. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση, να μειώσουμε την έκθεση και να αποφύγουμε τις σχετικές ασθένειες με τους καρκινικούς όγκους. Ε, η κατάργηση των φαρμάκων αυτών των τοξικών ε, και η αντικατάσταση από ε, μια λιγότερο επικίνδυνη ουσία δεν είναι κάτι εύκολο και εφικτό τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα κλειστό σύστημα για την παραγωγή, χρήση και απόσυρση των φαρμάκων. Τα κλειστά συστήματα στον τομέα της υγείας είναι επιτυχημένα ε, για την απομόνωση του κινδύνου, αλλά δεν χρησιμοποιούνται από την αρχή μέχρι το τέλος, χρησιμοποιούνται μόνο εν μέρη στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας των φαρμάκων σε ελεγχόμενο χώρο, σε φαρμακεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στα νέα αυτά στοιχεία κατασκευής των φαρμάκων, κλειστά στοιχεία, ε, κλειστές μέθοδοι, που θα προστατεύουν αυτούς που εκτίθενται περισσότερο, τους τεχνικούς και τους εργαζομένους και στις μεταφορές των αποβλήτων ε, όπου εκτίθενται όλοι όσοι εργάζονται στη μεταφορά των ουσιών αυτών. Συνεπώς λοιπόν αυτά προτείνω στην έκθεσή μου και όπως και στις προηγούμενες δύο οδηγίες είμαι διαθέσιμη <clears throat> να συνεργαστώ έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό ε, πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα στο σκιώδη συγγητή του ΕΛΚ. Α, λέγοντας ότι χαίρομαι που αυτή η τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων επιτέλους υπευλήθη για τις πρώτες δύο δέσμες ε, είχαμε συγκεκριμένη θέση, ιδιαίτερα για τη, τη δεύτερη δέσμη είπαμε ότι ε, επιστρεφόμαστε σε μία μόνιμη διαδικασία αναθεώρησης. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης χαίρομαι που εφαρμόζουμε μία μέθοδο που εδράζεται στη γνώμη των κοινωνικών εταίρων για το θέμα αυτό. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εύστοχο και σωστό. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμισμό που δείξαμε στις πρώτες δύο δέσμες ε, με ζητούμενο την συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσουμε γρήγορα στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω αμέσως ε, ότι εγώ θα ήθελα να διεκπαιρεώσουμε και την τρίτη δέσμη στη δική μας κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί προβλέπεται και τέταρτη δέσμη για το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διεκπαιρεώσουμε την τρίτη δέσμη ε, στη δική μας θητεία. Κάποια στοιχεία επιμέρους για αυτό το θέμα, παρόλο που η έκθεση θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε αυτή πρόοδο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα συγκεκριμένων κλάδων, συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δεχτούμε, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορούμε να δεχτούμε διαφοροποιημένη προστασία ανάλογα με το είδος του εργαζομένου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ε, ε, βοήθειας και στήριξης ε, και να λάβουμε υπόψη ε, τι ε, ιδιαιτερότητε των κλάδων. Σε ό,τι αφορά τα κύτταρο-τοξικά προϊόντα, έχω κάποιε επιφυλάξει. Όχι ω προ το εύρο ε, του ζητήματο, που είναι μεγάλο και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε λύσει για αυτά τα κύτταρο-τοξικά προϊόντα. Αλλά φοβάμαι ότι παρά είναι περίπλοκο και πολυθύτετο το θέμα για να το εντάξουμε και να το επιλύσουμε σε αυτό το θέμα. Αν και θα πρέπει να μα προβληματίσει. Επίση, τι εργαλεία έχουμε θα μας επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των ουσιών. Και τέλος μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά σας προειδοποιώ για να το ξέρετε, ε, στις τροπολογίες μου θα ξανακαταθέσω ε, κάποιες τροπολογίες για τις αναθυμιάσεις από τους κινητήρες, από τους διζελοκινητήρες και στον τριμερή διάλογο που θα έχουμε με την Αυστριακή Προεδρία, ε, το κάναμε και για, το δεύτερο, για τη δεύτερη δέσμη, ε, σας το λέω ότι αν ε, δεν καταφέρουμε να το επιλύσουμε στη δεύτερη δέσμη, θα ξανακαταθέσω τις ίδιες τροπολογίες στην τρίτη δέσμη μέτρων. Και συνεχίζουμε με το σκιώδη εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της κυρία Μαρίτα Ουρσκόγκ ζητώ συγγνώμη γιατί ε, ήθελα να έρθει αλλά είχε πρόβληματα χθε με την πτήση τη και γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, θα ήθελα η κυρία Ουρσκόγκ να ευχαριστήσει την κυρία Λαουραγκέα, την εισηγήτρια για την έκθεσή τη. Και να πω ότι η Μαρίτα πιστεύει ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ αξιόλογη και κατά τη γνώμη της δεν χρειάζονται αλλαγές ε, γιατί στηρίχθηκε στι συστάσει και τι συμφωνίε των κοινωνικών εταίρων η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τη κυρία Ατζέ για το κάδμιο και το Βιρίλιο ε, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο η κυρία Ουρσκόπ για να συνεννοηθεί με του επιστήμονε, του ερευνητέ και του κοινωνικού εταίρου. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τη ε, εισηγήτρια για τα υπόλοιπα, τα κυταρατοξικά φάρμακα. Φυσικά ε, και εμείς προβληματιζόμαστε για την υγεία των ε, εργαζομένων, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και την έκθεσή τους στα επικίνδυνα φάρμακα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε την έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκύψει θέμα αυτό, αλλά με προβληματίζει η πρόταση ήδη σε αυτό το στάδιο να, μπει στο παράρτημα, να μπουν στο παράρτημα ένα πολλά φάρμακα γιατί ούτε η επιστήμη ούτε οι κοινωνικοί εταίροι δεν είχαν την ευκαιρία να ε, εξετάσουν αυτές τις προτάσεις. Εξέτασε το κατάλογο φαρμάκων που ζήτησε η να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Για παράδειγμα, προτείνεται ε, στον κατάλογο ουσιών της οδηγίας ε, να συμπεριληφθούν ε, στρογόνα, προγεστερόνη ε, ή ε, συνδυασμός εστρογόνων και προγεστερόλης που χρησιμοποιούνται και για φάρμακα ελέγχου. Και αν συμπεριληφθούν αυτά τα φάρμακα στην νομοθεσία και καλυφθούν από την οδηγία, ουσιαστικά θα περιοριστεί η πρόσβαση των γυναικών στα φάρμακα αυτά σε όλη την Ευρώπη και κυρίως για αντισυλληπτικό σκοπό μια και θα χρειαστεί τέτοια ειδική διαδικασία για την νομοθεσία αυτή. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι απαράδεκτο. Τα φάρμακα του παραρτήματος 1 καλύπτονται, α, εμπίπτουν σε όλα τα άρθρα της οδηγίας και κυρίως το άρθρο 4.1 της οδηγίας που ζητά α, δυνατότητα υποκατάστασης. Αυτό μου σημαίνει ότι η πρώτη υποχρέωση του εργοδότη είναι, χωρίς να εξετάσει άλλους παράγοντες, να αντικαταστήσει αυτές τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Αυτό είναι πολύ αυστηρή διάταξη λόγω της φύσης αυτών των δραστικών ουσιών. Και μάλιστα αυτός ο κανονισμός είναι ο πιο αυστηρός που έχουμε στον τομέα της υγείας ε, και προστασίας. Η Μαρίτα θα αντιταχθεί στις προτάσεις που αποδυναμώνουν τις ε, διατάξεις οδηγίες ιδιαίτερα όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο αυστηρή τη διαδικασία στην πρώτη δέσμη. Θα πρέπει να δούμε μεμονωμένα, πιστεύει η Μαρίτα, κάθε φάρμακο ξεχωριστά, όπως έχουμε κάνει με όλε τι άλλες ουσίες μέχρι στιγμής. Και αυτή η διαδικασία θα πρέπει ε, να γίνει σε έναν επαρκή ε, χρόνο, γιατί η συμπερίληψη των φαρμάκων στην οδηγία αυτή ε, θα έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες. Οπότε θα μπορούσαμε, ακόμη και αν δεν τις περιελάβουμε στη συγκεκριμένη οδηγία, να εξετάσουμε άλλες ε, εναλλακτικέ λύσεις. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλή επιτυχία εφάρμοσε αυτή την προσέγγιση και πολλές ουσίες που ζητήσαμε στην πρώτη δέσμη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν περάσει τώρα στην τρίτη δέσμη, στην τρίτη φάση. Επίσης, ε, ζητάτε φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις, ε, από τα κράτη-μέλη προς τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία. Δεν συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Τα κράτη-μέλη μπορούν οικειοθελώς να ε, επιβάλλουν ε, φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά δεν μπορούμε να τα υποχρεώσουμε να το κάνουν. Σε ό,τι αφορά το πιθανά και το ενδεχομένως, probably και possibly, είναι προβληματική διατύπωση σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη κάποιων ρωσιών. Θα δημιουργήσει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Μία οδηγία είτε είναι, εντάσσεται, εμπίπτει στην οδηγία είτε όχι. Δεν μπορούμε να λέμε πιθανώς ή ενδεχομένως. Και μια και η Μαρίτα είναι και πρόεδρος, θα ήθελα να επισημάνει ένα μείζον διαδικαστικό θέμα. Λόγω της πρότασης για τα επικίνδυνα φάρμακα στην εργασία θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στα θέματα αυτά. Γιατί η δημόσια υγεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν ε, ρητή αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, οπότε θα πρέπει να αναμίξουμε πολύ πιο έντονα και αυτή την Επιτροπή. Κυρία Μακιντάιρ από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω γενικώ την τρίτη αυτή φάση του CMD και ευχαριστώ την εισηγήτρια που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Είπαμε και προηγουμένω ότι τα, οι ωριακέ τιμέ ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το αποτέλεσμα πολύχρονη διεξοδική ε, εξέταση, ε, αξιολόγηση και ελέγχων. Και μάλιστα έχουν πολύ αυστηρή διαδικασία για τη θέσπιση των οριακών τιμών. Οπότε δεν μπορούμε αυθαίρετα να αλλάζουμε το αποτέλεσμα μιας τόσο επίπονη προσπάθεια. Άλλωστε, ο απότερο σκοπό είναι να καταλήξουμε στι χαμηλότερε δυνατέ οριακέ τιμέ, ακόμη και χαμηλότερε από αυτέ που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ενεργά να επενδύουν στην επιστήμη και να ενθαρρύνουν τι εταιρείε και τι επιχειρήσει να επιδιώκουν τι χαμηλότερε δυνατέ ε, τιμέ και επίπεδα. Αλλά δεν θα πρέπει αυθαίρετα να ορίζουμε τόσο χαμηλά όρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν ε, ή να τα επιβάλλουμε, γιατί η ικανότητα εφαρμογής αυτών των ορίων στο χώρο εργασίας είναι το πιο σημαντικό. Ε, που το δεύτερο CMD δεν συμπεριληφθήκε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, γιατί από ξέρω η δεύτερη φάση του CMD εμπίπτει στι ε, διοργανικέ διαπραγματεύσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαπραγμάτευση για, το δεύτερο, για τη δεύτερη φάση, για τη δεύτερη δέσμη του CMD. Και τώρα μια πιο γενική παρατήρηση. Άσχετα με το τι θέλουμε να μπει στην τρίτη φάση του CMD, έχουμε εμ, πασχίσει για μια συνεκτική συνεπή διαδικασία. Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση του CMD. Αυτά που μάθαμε και συμπεριλάβαμε στις διαπραγματεύσεις μας καθοδήγησαν και στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων και θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα να διεκπαιρεώσουμε πλήρως τη δεύτερη φάση με ή χωρίς τον δίζελ, τις αναθυμιάσεις από τους διζελοκινητήρες. Ο κύριος Ρολά ε, εξέφρασε τη σχετική ανησυχία και μετά να περάσουμε στην τρίτη φάση του CMD. Ε, δεν λυπάμαι που ξεκινάμε τη διαδικασία, αλλά πρώτα πιστεύω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη φάση για να περάσουμε στην επόμενη, γιατί έχουμε μάθει πολλά από τη πρώτη φάση, έχουμε αλλάξει τη μεθοδολογία μας, έχουμε διδαχθεί από κάποια λάθη. Οπότε, αν έχουμε όλες τις διαδικασίες εκ παραλλήλου και όχι διαδοχικά όπως αρχικά είχαμε ξεκινήσει, πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Καλώς ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα πρέπει να αποκρισταλώσουμε τη θέση μας αν προηγουμένως δεν ολοκληρώσουμε τη δεύτερη φάση του CMD. Τώρα, για επιμέρους σημεία. Σημερίζομαι τον προβληματισμό σας για το πώς θα ε, μετρήσουμε την έκθεση στο κάδμιο συγκεκριμένα. Εγώ συμφωνώ με την εισηγήτρια που ζήτησε και εξέταση ουρών για να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, προστασία των εργαζομένων, γιατί μου είπαν ότι μόνο με καταμέτρηση της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε κάδμιο δεν αρκεί για να διαμορφώσουμε γνώμη. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και εξέταση ούρων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε και αυτή την εξέταση στην πρότασή της. Επίσης κάποιες εταιρείε και επιχειρήσεις εξέτασαν την πρόταση και εξέφρασαν προβληματισμό όχι μόνο για το κάδμιο, αλλά και για το βυρίλο και τη φορμαλδεΐδη. Και μάλιστα στην πατρίδα μου επιλήθηκε και το Αρμόδιο Συμβούλιο για την Υγεία και την Ασφάλεια. Μήπως λοιπόν και εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσουμε από, την, ε, από το Τμήμα Μελετών, το EPRS, να εξετάσει τη μελέτη αντικτύπου που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι μόνο για το βίριλο και τη φορμαλδεϊδή, αλλά και για άλλες ουσίες. Και κυρίως για το κάδμιο. Διερωτώμε αν θα μπορούσαμε και εμείς, η ε, υπηρεσία IPRS, να εξετάσει την ειδική μελέτη επιπτώσεων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τον τριμερή διάλογο, το είπαμε τον Ιούνιο, είμαι σε επαφή με την Αυστριακή Προεδρία και μάλλον θα ακολουθεί στο συντομότερο δυνατό, το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, μια ακόμη συνεδρίαση στο επίπεδο του τριμερούς διαλόγου, ο κύριος Καλβέτ Σαμπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα μιλήσω τώρα τη γλώσσα του Θερβάντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το κείμενο, το τρίτο στάδιο, η φάση μιας μόνιμης ε, επίθεσης ε, της Κομισιόνα και ημών όλων, όπως είπαμε, για την προσαρμογή, τη συνεχή προσαρμογή των επιπέδων, ε, ή μάλλον της μείωσης των επιπέδων κινδύνου ή έκθεση των εργαζομένων σε ορισμένου κατά την εργασία τους, είναι κάτι και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είναι μόνιμο εμείς που εργαζόμαστε το γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να έχει σχέση με την πρόθεση τεχνολογίας και των δυνατοτήτων μέτρησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως είναι προφανές, πολλές φορές μέγιστη προστασία έχουμε όταν υπάρχει μηδενική έκθεση. Το θέμα είναι όμως πώς μετράται αυτό η μηδενική έκθεση. Είναι μια μόνιμη προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι για το ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί. Μας ικανοποιεί η προσέγγιση της Κομισιόν, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και το έργο της εισηγητριάς μας και η προσέγγισή της. Και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Απλά πρέπει να έχουμε κατά το τέλειο είναι εχθρός του καλού. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος ε, και όπως θέλει και η κυρία Αγκαία θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, δώσουμε πρόοδο και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Έχουμε συσσωρεύσει εμπειρία στο πλαίσιο της εξεργασίας των δύο πρώτων δεσμών. Η φιλοδοξία μας λοιπόν δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προσκόμματα στην πρακτική εφαρμογή σε ό,τι αφορά το ντίζελ ε, στη δεύτερη ε, δέσμη. Εγώ είχα ψηφίσει και είχα συμμετάσχει και συμφωνώ να περιληφθεί το δίζελ. Είχα εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη μου τότε και ισχύει αυτό που πίστευα τότε. Όμως ε, δεν θέλω να υπάρξει πρόσκομα εξ αυτού, να υπάρξει αδιέξοδο και έτσι να καθυστερήσουν οι υποφελείς συνεπές για τους εργαζομένους. Οπότε ε, πρέπει να αποφύγουμε να μπλοκάρουμε και την τρίτη δέσμη. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρακτική εφαρμογή. Στηρίζω όπως είπα για τον ντίζελ τις προτάσεις, όμως ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τον πιο γρήγορα. Ε, για πιο τεχνικές πτυχές της έκθεσης τώρα. Συνολικά στηρίζω τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου και για το κάδμιο συγκεκριμένα. Για τις πιο τεχνικές πτυχές πρέπει να πω ότι μαθαίνουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι ε, ειδικοί επί του θέματος όπως η Μαρίτα που έχει αυτή την τύχη. Μαθαίνουμε ακούγοντας, διαβάζοντας ε, και ακούγοντας συγκεκριμένα τους κοινωνικούς εταίρους. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε την πρόταση οδηγία που είναι ήδη καλή. Για τα κοιτοτοξικά και για τα φάρμακα. Δεν μας ε, ε το, το σημαντικό δεν είναι ο συγκεκριμένο ε, ανθρακορίχο ή τεχνικός εργαστηρίου, αλλά το εργαστήριο, για παράδειγμα, ο χώρο που εκτίθεται. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε στον δυνατόν ε, μεγαλύτερες εγγύησεις. Και έχοντας υπόψη πιο πολύ και τις οικονομικές παραμέτρους, αλλά τις πρακτικές και πολιτικές για να μην ε, υπάρξει εμπλοκή όπως είπε και η κυρία Μακιντάιρ, γιατί θέλουμε να κλείνουμε ε, τα στάδια, να μην αφήσουμε και τα τρία ανοιχτά, για παράδειγμα, στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων. Τέλος. Κυρία Αγκαία, Φυσικά θα δει όλες αυτές τις οικονομικές πτυχές, οικονομική σκοπιμότητα και για τις ΜΜΕ νομίζω ότι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα προσεγγίζει το θέμα και θα αναλύσουμε και εμείς ε, τις ε, προτάσεις της ε, ευνοϊκά διακείμενη προς αυτές. Γιατί ο στόχος είναι να προσφέρουμε πραγματική βοήθεια και μέτρα που θα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βελτιώσουν την προστασία όχι να κρύβουν, ε, να προσπαθούν να συγκαλύπτουν τα πράγματα. Θα εργαστούμε λοιπόν με την καλύτερη δυνατή διάθεση και πνεύμα και προσυπογράφω όλα όσα έχουν υποθεί και ε, γραφεί, γιατί νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική βάση αν θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, Θέλω να χαιρετήσω τη συνάδελφο Λάουρα για το έργο της στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης ε, για την περιορισμό της έκθεσης ε, σε καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους ε, παράγοντες ή ουσίες. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων θα ήθελε να υπάρχουν νέα όρια έκθεσης για 50 ουσίες μέχρι το 2020. Άρα έχουμε μπροστά μας ακόμη πολλή δουλειά. Φυσικά δική μας ευθύνη και δικός μας ρόλος είναι να εργαστούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ανεξαιρέτως την προστασία για όλους τους εργαζομένους ε, σε ό,τι αφορά τα, το τοξικά, τα τοξικά φάρμακα. Ε, είναι φάρμακα χρήσιμα γιατί τα καρκινικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ε, νόσων που προ που προκαλούνται από την υπερβολική έκθεση ε, σε κάποιε ουσίες είναι κάτι που μα απασχολεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τους νοσηλευτές, ε, που χειρίζονται στι ουσίες και είναι εκτεθειμένες πολλές φορές αυτού του κινδύνου. Είναι δηλαδή ουσιαστικά δηλητήρια τα φάρμακα αυτά για ορισμένου εργαζομένου. Και αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα πρωτόκολλα χρήση αυτών των φαρμάκων να ε, ενισχυθούν, να δούμε αντίστοιχα αποτελέσματα κλινικών μελετών και να περιορίσουμε τη διάρκεια έκθεσης. Η πρόταση για καθορισμό των ορίων έκθεσης 8 ε, ώρες τη μέρα, 40 ώρες την εβδομάδα, είναι μια χρήσιμη διάταξη, είναι ένα όριο που βάζουμε, διότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό Δυστυχώ πολλέ φορέ εργάστηκε περισσότερε ώρε, άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι με τι ε, περορίε που ενδεχομένω εργάζονται εκτίθενται για περισσότερε ώρε αυτού του ε, δυνητικού ε, καρκινογόνου παράγοντε. Υπάρχει και η πρόταση για τη στήριξη οικονομική, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό. Είναι Μια πρόταση που μπορούμε να στηρίξουμε, όμω δεν θα πρέπει να μα διαφύγει το ουσιώδε που είναι η προστασία τη υγεία των εργαζομένων. Εξού και έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την πρόταση ε, παράτασης ε, του χρόνου προσαρμογής ε, από 5 σε 7 έτη και δική μας ευθύνη είναι η πρόληψη των κινδύνων. Πρέπει να δώσουμε βέβαια τη δυνατότητα να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη. Υπάρχουν ιατροί υγείας που προτείνουν διάφορα μέτρα και θέλουμε να περιορίσουμε την έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Στηρίζω την πρόταση που έκανε πριν ο πρόεδρός μας, δηλαδή να μην Μα διαφύγει σημασία που έχει να επανακατατεθούν ε, οι τροπολογίε ε, για την έκθεση σε καυσαέρια ε, από χήματα που καίνε είναι Είναι κάτι που ενδιαφέρει και την κοινή γνώμη, ένα θέμα πολύ σημαντικό, διότι αφορά, θίγει πολλού συμπολίτε μα. και εργαζομένους. Δεν υπάρχει ε, τιμή ε, για την υγεία. Κυρία Ντέλη, ο πρόεδρος δεν είναι εδώ και δεν βλέπω και ένα άλλο συνάδελφο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Όλσεν ευθύς αμέσως από την πλευρά της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για μια εξαιρετική έκθεση. Είναι, είναι ικανοποιητικό για μας να παρακολουθούμε τη συζήτηση αυτή όταν βλέπουμε το τι γνώση και κατανόηση υπάρχει. Θα ήθελα να κάνω 7 πάρα πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχει ήδη τεθεί, ότι πρόκειται για μια φανταστική οδηγία. Είναι μια πολύ ισχυρή οδηγία. Όταν μια ουσία εντάσσεται στην οδηγία υπάρχει αυτόματο αίτημα αντικατάστασης και δεν περιορίζεται το αίτημα αυτό από τεχνικά ε, όρια. Δεν υπάρχουν οικονομικές επίσης ε, μορφές περιορισμού. Συνεπώς λοιπόν αυτή τη στιγμή η οδηγία αυτή, η ουσία στην οδηγία, ε, οφείλουμε να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε μια τόσο επιστημονική και αυστηρή διαδικασία για την ένταξη. Έχουμε τον τριμερή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, έχουμε μια μελέτη επιπτώσεων και έχουμε φυσικά και τους συνομοθέτες. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο γρήγορα όσο κάποιοι θα το επιθυμούσαν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται σε αυτό το οποίο ήδη εσείς έχετε αναφέρει, Πρόεδρε, στην ανάγκη δηλαδή η ενημέρωση της οδηγίας αυτής να γίνει μια τακτική διαδικασία απολύτως αποδεκτή. Η Επίτροπος Τίσεν και ο Πρόεδρο Ιούνκια έχουν υποστηρίξει την πρόταση αυτή, θεωρούν ότι είναι σημαντικό στοιχείο του κοινωνικού πυλώνα και κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της διαδικασίας αυτής. Ε, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση, στην πέμπτη φάση, στην έκτη φάση, αλλά χρειάζεται χρόνος για να το κάνουμε με σωστό τρόπο. Είναι λοιπόν σημαντικό η δεύτερη και η τρίτη φάση να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό είναι πολιτική ευθύνη και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω ότι το Συμβούλιο μέχρι τώρα ήταν θετικό στις προτάσεις της Επιτροπής και πιο γρήγορα από όλους τους άλλους τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Ένα τρίτο σημείο συνδέεται με τα δύο προηγούμενα και αφορά τα κυταροτοξικά φάρμακα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Η Επίτροπος είναι η ίδια εμπλέκεται και βασικός μας στόχος είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε εφικτές λύσεις για να βοηθήσουμε τα 12 εκατομμύρια εργαζομένων στους οποίους αναφέρθηκε η συγγήτρια. Αυτό περιλαμβάνεται έτσι και αλλιώς στην οδηγία πλαίσιο, γενικά για την υγεία, στον τομέα της εργασίας. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθούμε και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Όμως, όπως ήδη υπόθηκε, το να βάλουμε μία ομάδα φαρμάκων στην οδηγία αυτή δημιουργεί και κάποιες σοβαρές νομικές και πολιτικές ε, πλευρές. Δεν προσπαθούμε απλά να διατητεύσουμε απλά μέσα στα κέρδη των επιχειρήσεων και το συμφέρον των εργαζομένων, την προστασία των εργαζομένων. Μιλάμε για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα της φροντίδας και της προστασίας. Εδώ η νομική μας υπηρεσία το ψάχνει ακόμα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία φαίνονται στην έκθεση, το πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια σημεία κρίσης μέσα στην οδηγία αυτή. Είναι μια αυτόματη οδηγία Υπάρχει δηλαδή μια αξιολόγηση, αν υπάρχει μια αξιολόγηση που λέει ότι η αποτελεσματικότητα της φροντίδας είναι τέτοια δύσκολη και ακριβή που θα μπορούσε να μας οδηγήσει απευθείας στη διαδικασία αντικατάστασης. Αυτό είναι περίπλοκο και είναι και κάτι το οποίο πολιτικά και οικονομικά πρέπει να μελετηθεί σοβαρά. Ευχαριστώ πρόεδρε. η κυρία Τζέα. Να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, απόψεις τις οποίες εξέθεσε. Είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να εργαστούμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Πρόκειται για μια βάση βελτιώσιμη με τη συμμετοχή των πάντων. Υπάρχουν κάποιες απορίες σε σχέση με τα λεγόμενα επικίνδυνης χρήσης φάρμακα. Μιλάμε για την αντικατάσταση θεραπείων που σώζουν τη ζωή εκατομμυρίων ίσως ασθενών. Ζητάμε λοιπόν οι διαδικασίες και οι φάσεις ε, ε, προετοιμασίας και προπαρασκευής των φάρμακων να γίνονται με προστατευόμενο τρόπο έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα φάρμακα αυτά που σώζουν ζωές και για τα οποία δεν υπάρχουν αντικατάστατα αυτή τη στιγμή να γίνεται η παρασκευή των φαρμάκων αυτών, των ουσιών αυτών με ασφαλή τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι δίνουμε μια σωστή κατεύθυνση εγώ δεν θέλησα να μειώσω ακόμα περισσότερο τα όρια. Νομίζω ότι βασικός στόχος, όλοι το ε, μοιραζόμαστε αυτό, είναι να καταργήσουμε τις, καρκινο, ε, τις ουσίες που προκαλούν καρκίνο, τις καρκινογόνες ουσίες. Θα πρέπει στα πλαίσια της μεταβατικής φάσης να βρούμε και νέες ουσίες, νέα υλικά, νέα φάρμακα, που να προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν Ίσως η μεταβατική περίοδος αν μεγαλώσει λίγο είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις να μην κλείσουν. Η επιλογή μας λοιπόν ως ε, συνομοθέτες είναι σαφής. Το είπε και ο κύριος Λέιαρικ, η υγεία των εργαζομένων δεν έχει τίμημα. Αν ε, βέβαια χαθεί η θέση εργασίας γιατί πρέπει να φύγει, να πάει αλλού η επιχείρηση ή να κλείσει η επιχείρηση, Καλό θα είναι να προβλέψουμε μέσα στήριξης των εργαζομένων αυτών που θα χάσουν τη δουλειά τους. Στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτής της βάσης λοιπόν εργασίας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τους εκπροσώπους των εργαζομένων όπως επίσης και των βιομηχανιών. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο συμφέρον ή ενδιαφέρον προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Βασικό μου βασικός μου στόχος είναι η υγεία των εργαζομένων αλλά και η υγεία των επιχειρήσεων και η οικονομική ευημερία, χωρίς όμως να φύγεται η υγεία των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω λοιπόν το αίτημα να με βοηθήσετε να βελτιώσω την έκθεση αυτή. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια καλή βάση και μπορούμε να πετύχουμε κάτι θετικό στο τέλος. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ευγενείς κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Εξαιρετική και γενναία η δουλειά που έχει κάνει ιδίω σε ό,τι αφορά την έκθεση των εργαζομένων, των επαγγελματικών τομέα της υγεία στα κοιτάρτοξικά φάρμακα. Υπάρχει κίνδυνος, ε, υπάρχουν ε, επιβλαβείς συνέπειες από την χρόνια έκθεση, ε, τακμηριωμένη με στοιχεία εδώ και 30 χρόνια. Κάθε χρόνια χιλιάδες επαγγελματίες στο τομέα της υγείας πεθαίνουν από λευχαιμία, έχουν προβλήματα αναπαραγωγική υγεία, από βολές, δυσπλασίες κτλ. Ε, κτλ. Ε, μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις για τους επαγγελματές υγείας. Ε, λίγα φάρμακα περιλαμβάνονται στις αλλά τα πιο πολλά καρκινογόνα όπως ορίζονται από το ΙΑΡΚ. και στο παράρτημα 1. Για τα επίπεδα έκθεσης, στον χώρο εργασίας. Ε, εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε ίσως ακριβώς ε, τα ε, ποσοστά, τα νούμερα των εργαζομένων που εκτίθενται. Υπάρχουν, όπως είπα, στοιχεία εδώ και χρόνια. Ε, μπορούμε να κάνουμε όμως, αν υπάρχει βούληση και στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης, μια μελέτη αντικτύπου. Είναι τροπολογίες αυτές που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά ε, εθνικά συνδικάτα, από τους κοινωνικούς εταίρους, από τους φαρμακοποιούς, από τους νοσηλευτές, από ακαδημαϊκούς. Όλοι ε, συμφωνούν γιατί τους έχουμε συνομιλήσει και όλοι θέλουν δράση να αναλυφθεί τώρα και όχι κάποια στιγμή ε, από μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τώρα. Ε, οι τροπολογίε που έγιναν στο πλαίσιο τη δεύτερη δέσμη θέλουν να, επίσης να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και υπάρχει δέσμευση για κατάθεση νέων τροπολογιών στο πλαίσιο της τρίτης φάση. Δεν κατάφερε να καταθέσει προτάσει η Κομισιό για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Το μόνο που κάνει είναι επαναλαμβάνει ότι έχει εκδώσει κατευθυντήριε γραμμέ. Πότε έγινε όμω αυτό, το 2010. Πρέπει επομένω να υπάρξει επικαιροποίηση τώρα, εφόσον έχουμε τεχνολογικέ εξελίξει που το καθιστούν αναγκαίο. Και τελικά η καθοδήγηση τη Κομισιόν δεν είναι παρά κάτι που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αλλά εμεί θέλουμε να υπάρχει πραγματικό αντίκτυπο, άρα θέλουμε νομοθεσία. Και υπάρχει κίνδυνο, αν δεν αναλυφθεί τώρα δράση, η Κομισιόν να μην μπορέσει σε δύο χρόνια ή τέσσερα χρόνια ή δέκα χρόνια να αναλάβει δράση και να είμαστε ε, μετά από μια δεκαετία ξανά εδώ να καθόμαστε και να λέμε όλοι πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και μόνο ο εισηγητής όμως να λέει τι θα γίνει τώρα. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 4 Σεπτεμβρίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 24 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 18 Οκτωβρίου. Πέραμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Εξέταση ε, ε, σχεδίου ετήσιας έκθεσης για την ε, απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωζώνη. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο για 10 λεπτά στον κύριο Σφεν Λάγκεντεκ και λυπάμαι αν δεν το πρόφερα σωστά το όνομά σας, που είναι τμήματάρχη στο Κοινό Κέντρο Ερευνών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνατε να σας παρουσιάσουμε τον πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων ευκαιρία της ετήσιας έκθεσης μας. Το περασμένο Νοέμβριο οι ηγέτες ε, στην κοινωνική διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμπορκ επέβαλαν τις, προ... τις ε, δεσμεύσεις τους για 20 θεμελιώδεις αρχές και αξίες που ε, απαιτούνταν για εύρυθμες αγορές εργασίας και εργασιακά συστήματα. Ο πρόεδρος Ιούγκερ είπε από το δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς, ε, σε υγειονομική περίθαλψη, σε διασμό επαγγελματικής ιδιωτικής ζωής ε, και ένα ελάχιστο κοινωνικό πυλώνα, ε, ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να προσαρμοστούμε στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Και μάλιστα στο χειμερινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την, με την εξέταση πρόοδου σε κοινωνικές και άλλες προτεραιότητες έχουμε δει τις, ε, το βαθμό εφαρμογής των συστάσεων αναχώρα και για πρώτη φορά οι διάφορες εκθέσεις αναχώρα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τα στοιχεία από τον πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων ε, συμπεριλήφθηκαν στην παρακολούθηση των κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών. Ο πυρώνας εντάσσεται στην, ε, γενική, στο γενικό κοινωνικο-οικονομικό θεματολόγιο της Επιτροπής, ε, προκειμένου να βελτιωθούν οι βιωτικές και εργασιακές συνθήκες. Ε, θέλουμε ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δυναμικές αγορές εργασίας, δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δημόσια υποστήριξη, κοινωνική προστασία και ένταξη. Επίσης αυτές οι τρεις διαστάσεις καλύπτουν 12 ε, τομείς. Έχουμε 14 δείκτες και 21 δευτερογενείς επικουρικούς δείκτες στον πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων. Επίσης έχουμε ταξινόμηση ανά φύλλο εκπαίδευση και έχουμε 93 τέτοιους, 93 ε, επιμέρους δείκτες με βάση τις πηγές της Eurostat, του ΟΣΑ και άλλων ε, ερευνών και μελετών. Το επιτελείο μας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, παρακολούθησε αυτή την ανάπτυξη δικτών ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια στατιστική συνοχή τους και έχουμε και μάλιστα σε 24 γλώσσες ε, ένα τρόπο ανάγνωσης επιγραμμικό. Βλέπετε στο link και μπορείτε να το βρείτε χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης και σημειώνοντας το Social Scoreboard, το πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων, που μας δίνει πολλές πληροφορίες, τις οποίες ε, ε, ταξινομήσαμε σε έξι είδη γραφικών παραστάσεων που είναι interactive. Έχουμε ένα για την, για την κοινωτική σύγκληση, για τις κοινωνικές προκλήσεις, κοινωνική σύγκληση και το πρώτο είναι social granularity. Βλέπουμε ποια είναι η προσθέμενη αξία της αναλυτικής ε, ε, ταξινόμησης των διαφορών στοιχείων αναομάδων πληθυσμού. Βλέπετε εδώ το παράδειγμα των ε, ποσοστών απασχόλησης, για παράδειγμα. και μάλιστα έχουμε από 57,8% στην Ελλάδα και 81,8% στη Σουηδία ποσοστό απασχόλησης. Επίσης, ε, ε, με, την, με τα αναλυτικά στοιχεία έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ε, έχουμε και στοιχεία ανά φύλλο. Βλέπετε ότι στη Σουηδία, Λιθουανία, και κάποιε άλλε χώρε τα ποσοστά απασχόληση είναι παρόμοια σε άντρε και γυναίκε. Ενώ σε άλλε χώρε μέλη, Μάλτα, Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία για παράδειγμα, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ στην απασχόληση ανδρών και γυναικών. Έτσι έχουμε ε, πληροφορίε και μπορούμε να κατευθύνουμε καλύτερα τι πολιτικέ απασχόληση. Άλλο διαχωρισμό ε, είναι με βάση την ηλικία. Έτσι βλέπουμε καλύτερα που επικεντρώνονται οι προκλήσεις για διάφορες ηλικιακέ ομάδες, πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους ή νέους εργαζόμενους. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, έχουμε για τους νέους υψηλά ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα από τις άλλες χώρες. Και βλέπουμε τις ιδιαίτερες προκλήσεις και για τους ε, πολύ νέους εργαζόμενους και για τους πιο ηλικιωμένους. Άλλη, ε, άλλος διαχωρισμός γίνεται με βάση τις ε, το μορφωτικό επίπεδο. Βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μισό εργατικό δυναμικό με ε, χαμηλή δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι άνεργο. Και βλέπουμε το χάσμα μεταξύ των ε, λιγότερο μερφωμένων και περισσότερο μερφωμένων να είναι πολύ μικρό στην Πορτογαλία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και περνάμε στο δεύτερο βαθμό ε, πληροφοριών στο δεύτερο πίνακα που αφορά την σύγκληση, την κοινωνική σύγκληση. Ο πυλώνας αυτός ε, γίνεται η πηξίδα ε, για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση και την ε, επίτευξη καλύτερων βιωτικών συνθήκων και εργασιακών συνθήκων, ώστε να έχουμε μια κούρσα προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και μάλιστα αυτά, αυτές οι γραφικές και χρονικές απεικονίσεις μας δίνουν μία εικόνα για το κατά πόσο η σύγκληση γίνεται προς καλύτερες επιδόσεις με βάση αυτούς τους βασικούς δείκτες. Για παράδειγμα, εγκατάλειψη του σχολείου και έχουμε τις ε, διαφορές μεταξύ των καλύτερων και των χαμηλότερων επιδόσεων σε συγκεκριμένη χρονιά. Και έτσι, αν θέλουμε να μειώσουμε την εγκατάλειψη του σχολείου, εκεί βλέπουμε ότι το επιθυμητό είναι μία σύγκληση προς τα πάνω. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε ό,τι αφορά το εισόδημα και την ισότητα. Δεν υπάρχει τέτοια ε, επιθυμητή σύγκληση για τα επίπεδα ανεργίας επίσης. Και τώρα, αν με ρωτήσετε πόσους από τους 14 βασικούς στόχους δείχνουν μία σύγκληση προς τα πάνω, Αν ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους 14 βασικούς δείκτες, μόνο σε τρεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, σύγκληση προς τα πάνω. Στους υπόλοιπους ε, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε τέτοια σύγκληση. Και το τελευταίο είδος ε, γραφικών ε, απεικονίσεων, το εργαλείο που έχουμε, είναι κάποιοι χάρτες που δείχνουν που επικεντρώνονται οι συγκλήσεις οι βασικές προκλήσει για τις επιμέρους χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, heat map, όπως λέμε, που έχουμε τι τις βασικές επιδόσεις ε, στους ε, κύριους δείκτες. Και έχουμε πέντε χρώματα με 20% των ε, οριακών τιμών από 12 χρόνια παρατηρήσεων. Το MOV είναι οι καλύτερες επιδόσεις, το άνω 20%, καλύτερες τιμές και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει τα κράτη-μέλη από το 2005 μέχρι το 2015, βλέπετε το Βέλγιο που είναι αριστερά έχει τέσσερις, ε, ε, τέσσερα τέτοια μόβ τετραγωνίδια για την ε, ανισότητα, την βρεφονιπιακή φροντίδα, το εισόδημα. Βλέπουμε ότι εκεί έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις στο Βέλγιο. Βέβαια αυτό δεν δεν δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες το Κοινό Κέντρο Ερευνών εξέτασε διάφορους αλγόριθμους για την ε, ανακατανομή αυτών των χαρτών και βλέπουμε πού βρίσκονται οι περισσότερες προκλήσεις και σε ποιους δείκτες ε, οι χώρες αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις και οι χώρες στα δεξιά είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες προκλήσεις. Οπότε βλέπουμε το χάρτη αυτό για το 2016 ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της οι πιο επίγουσες προκλήσεις αφορούν την ανισότητα, εισοδηματική ανισότητα, αντίκτυπο των ε, κοινωνικών μεταφορών και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και ένδυας. Και όταν βλέπουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις αυτούς τους τομείς, βλέπουμε ότι είναι η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Λετωνία. Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται και με τις ε, έρευνες του τελευταίου Ευρωβαρομέτρου που δείχνουν ότι τα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα που προβληματίζουν τους πολίτες είναι η ανισότητα, η κοινωνική προστασία και η ανεργία. Βέβαια, αυτές οι προκλήσεις ήταν διαφορετικές το 2010. Εκεί η ε, μεγαλύτερη ανησυχία ήταν η, ήταν η ανεργία η σχολική εγκατάλειψη και η ανισότητα εμφανίστηκε αργότερα. Μάλιστα πριν την κρίση είχαμε ακόμη πιο διαφορετικές ε, ανησυχίες. Ήταν περισσότερο ε, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων, η σχολική εγκατάλειψη, οι διατάξεις ε, για την βρεφονιπιακή φροντίδα. Εν κατακλείδη, θέλουμε μια πιο συνεκτική Ευρώπη με περιορισμό των αποκλεισμών και με τις κοινωνικές επιδόσεις των κρατών μελών έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία για πιο ισορροπημένη διακυβέρνηση. Και μάλιστα το εργαλείο, το επιγραμμικό του πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων ε, μας ε, βοηθά να λάβουμε πιο εμπεριστατωμένες ε, αποφάσεις. Και μάλιστα το εργαλείο αυτό υπάρχει σε 24 γλώσσες, επικαιροποιείται άμεσα ανάλογα με, τις, με την ενημέρωση που κάνει και η Eurostat online και μάλιστα πολύ ευχαριστώ ε, να ακούσω τις προτάσεις και τις συστάσεις σας. Merci. Σας ευχαριστούμε. Για το ΕΛΚ, κύριε Χέτμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έκανε. Ε, και πιστεύω ότι θα εμπλουτίσει τη συζήτησή μας. Βέβαια, είναι να αναφυσβήτητο ότι πρώτη φορά φέτος η απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα ε, αποτέλεσαν το αντικείμενο ειδική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δική μα και δεν ήταν απλώς ε, η γνωμοδότηση που δίναμε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Ε, σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα και την απασχόληση, αυτό πια γίνεται σημαντικό τμήμα του συνόλου της οικονομική πολιτική και τη πολιτική συνοχή, Γι' αυτό και χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, αυτό είναι σημαντικό, ώστε με βάση τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα πολιτική συνοχή και κυρίω για, για το νέο ενισχυμένο κοινωνικό ταμείο, η νέα πολιτική συνοχή θα συνδέεται περισσότερο με τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για πολύ καιρό διαπιστώσαμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πραγματικά άρχισε να ανακάμπτει σε τομείς όπω τα δημόσια οικονομικά, η απασχόληση ή οι επενδύσει το επίπεδο ανεργίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του 2018 ήταν περίπου 9%, ούτε καν 9% και είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση. Θα ήθελα πάντως να υπογραμμίσω ότι αυτή η μείωση της ανεργίας δεν είναι αρκετή, ούτε μας ικανοποιεί ιδιαίτερως. Θα ήθελα στην έκθεσή μου να τονίσω μερικούς βασικούς τομείς ε, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για παράδειγμα, η ανεργία των νέων, η παραγωγικότητα, η αύξηση των μισθών, οι συντάξεις, η κοινωνική πρόνοια ή το σύστημα υγείας. Ε, χαίρομαι για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις στάσεις αναχώρα. Κατά τη γνώμη μου κάνουν πολύ καλή ανάλυση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και αποτελούν ε, σημαντικό αναπόσπαστο στοιχείο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ταυτόχρονα αυτό που μας ανησυχεί είναι ο χαμηλός βαθμός εφαρμογής των συστάσεων αυτών από τα κράτη-μέλη. Αυτή η κατάσταση παρεμποδίζει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Βέβαια, εδώ έχουμε την, τις συστάσεις αναχώρα για τις χώρες Ευρωζώνης, αλλά δεν έχουμε κάποιες οικουμενικές συστάσεις καθολικές που ε, υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι βασικό μα στόχος θα πρέπει να είναι κυρίω ε, η δημιουργία μια ε, συνεκτική αγορά εργασία και να εξασφαλίσουμε υψηλό ποσοστό απασχόληση για όλου και κυρίω για τι πιο μειονεκτικέ ομάδε. Γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθούν αξιόπιστε συμβάσει εργασία και αποτελεσματική κοινωνική πρόνοια. Ε, κυρίως και για τις άτυπες μορφές ή τις νέες μορφές ε, συμβάσεων εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να λάβω υπόψη τις ραγδαία εξελισσόμενες θέσεις εργασίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα πρέπει να εφοδιάσουμε τους εργαζόμενους με νέες δεξιότητες και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διαβίου κατάρτιση. Επίσης να προωθήσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων και να επιτρέψουμε καλύτερη είσοδο και επανείσοδο στην αγορά εργασίας. Εν κατακλή θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη ε, πολιτική εξισορρόπησης του ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, ώστε να έχουμε ελαστικές ε, ημέρες εργασίας, καλύτερη αξιοποίηση της γονικής άδεια και εξασφάλιση καλύτερης ε, μέρημνας για τα παιδιά. Προσβλέπω σε πολύ επικοδομητική συζήτηση και σε καρποφόρα συνεργασία για την έκθεση αυτή. Και περιμένω τις προτάσεις και τις συστάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σκιώδης εισηγητές, ε, Χάβι ε, για του Σοσιαλιστέ Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας για τη δουλειά του, το σχέδιο έκθεση. Είναι πολύ καλό, το έχουμε λάβει. Ο σκιώδης εισηγητή για την ομάδα μου θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι μια καλή αφετηρία το έργο του εισηγητή για να εργαστούμε αυτές τις εβδομάδες τονίζει και περιλαμβάνει και το έργο το προηγούμενο της Κομισιόν ε, με τις ειδικές ε, αναχώρες συστάσεις και τις προτεραιότητες της Κομισιόν. Ε, Σημερίζομαι εν μέρη τα όσα αναφέρατε και τις ευαισθησίες σας και ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε στην ίδια γραμμή. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια όμως. Ο κίνδυνος που υπάρχει ο κίνδυνος που βλέπουμε εμείς να εφίσταται όταν μιλάμε για τις στάσεις αναχώρα, όχι τόσο σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του αλλά της ε, τη γενική κατάσταση και τις γενικές πατήσεις κομισιών για την οικονομική κατάσταση. Φοβούμαστε ότι υπάρχει κίνδυνος αυταρέσκειας. Τα μακροοικονομικά δεδομένα βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε τρεις πτυχές, κυρίως την ανάπτυξη, φυσικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και τη μείωση του ελλείμματος, εντάξει, και τη μακροοικονομική σταθερότητα των εθνικών προπολογισμών. Τρεις είναι οι βασικοί αυτοί δείκτες ε, που σημειώνουν ε, μεγάλη βελτίωση και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, επανερχόμεθα σε επίπεδα προ-οικονομικής κρίσης. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και σε θέση να ε, δείχνουμε ε, ότι υπάρχουν και κάποια τροτά ε, στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δύο κινδύνους που βλέπω. Τα τελευταία δέκα χρόνια βλέπουμε σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα να μην έχουμε την ανάκαμψη που θα θέλαμε και με μια μεγάλη διαφορά που έχουμε από σήμερα και πριν 10 χρόνια είναι ότι αυξήθηκε το χρέος σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό μας ε, δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Ε, πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και μια πιθανή μελλοντική κρίση. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί είπα να μην είμαστε και να δούμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αν υπήρξε αύξηση, αυτό βασίζεται σε αποφάσεις που λάβαμε αλλά και σε αποφάσεις που δεν λάβαμε. Οικονομική ανάκαμψη βασίζεται στην νομισματική πολιτική της ε, ΕΚΤ που είναι υπερεπεκτατική και σε κάποια θετική ε, ατμόσφαιρα ε, σε κάποιες χώρες με οικονομική ανάκαμψη, κάτι που δεν είναι σύνηθες, αλλά και με χαμηλές τιμές πετρελαίου. Και αυτό ωφελεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Όταν όμως ε, χαθούν κάποια από αυτά τα θετικά στοιχεία, θα είμαστε έτοιμοι, αυτό το ερώτημα. Θα είμαστε προετοιμασμένοι. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση που θα έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει. Και πρέπει να κάνουμε αρκετά πράγματα, επαρκή πράγματα από θεσμικής πλευράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ουσιώδεις αλλαγές ε, στις κοινωνίες μας, ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε μια δυνητική μελλοντική κρίση. με κάτι μας ανησυχεί Και παράλληλα πρέπει να κάνουμε και το απαραίτητο έργο ε, για να δούμε τι ε, πληγές, τι ουλές άφησαν οι πληγέ των τελευταίων ετών και πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις πληγές, ε, το μισθολογικό χάσμα, ε, συντάξεις, φτώχεια, νεανική ανεργία, μακροχρόνια ανεργία. Και επίσης υπάρχει και ένα εργαλείο που τα τελευταία τέσσερα χρόνια δούλεψε από αυτού ε, πολύ κομισιόν και μιλάω για τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι το εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα ο κοινωνικό πυλώνας, ε, για να κλείσουμε αυτές τις ε, πληγέ. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ηθικό, αλλά γιατί θα μας δημιουργήσει, θα μας βοηθήσει να έχουμε και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Για τα δύο, τελευταία, πολύ γρήγορα, ένας μεγάλος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Παραμένει πολιτικός κίνδυνος, το βλέπουμε παντού στον κόσμο και πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα που δρομολόγησε ο πρόεδρος Τραμπ. Πολύ μεγάλος ο πολιτικός κίνδυνος για την οικονομία και δεύτερο στοιχείο οι δημόσιε, μάλλον πολιτικές αρχές εμεί δεν αποφασίζουμε τον οικονομικό κύκλο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία αυτό όμως που εμείς αποφασίζουμε και αυτό που εξαρτάται από εμάς είναι πού θα επωφεληθούμε και πότε από τον κύκλο, όταν θα είναι στην επεκτατική του φάση, όπω τώρα, αν θα μπορέσουμε δηλαδή να αποφεληθούμε με θετικό τρόπο και όταν είναι σε αρνητικό επίπεδο, αν μπορούμε να προσβέσουμε τι επιπτώσει που θα έχει ο αρνητικό κύκλο. Και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε τώρα και αν τα πράξουμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. ECR, Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Μα έδειξε παρουσίαση της Κομισιόν, αλλά και τα αποτελέσματα που είχαμε ε, την Άνοιξη, ότι με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βλέπουμε πόσο μεγάλη ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ε, υπάρχει στο ε, επίπεδο το ευρωπαϊκό. Η προσέγγιση του εισηγητή είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και δείχνει και αυτή πόσο είναι πήγον να αναλυφθούν μεταρρυθμίσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη. Ε, όπως παραδείγματο χάρη ψηφιακά προσόντα και δεξιότητες, ε, ε, ένα σύστημα βιωσιμότητας. Προτείνουμε εμείς ως ECR ένα, μια δέσμη τροπολογιών για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και πιο βιώσιμη παραγωγικότητα βέβαια. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πρέπει να έχουμε υπόψη μα τη συνολική εικόνα και πραγματικά στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη σύγκληση. Ε, αυτή η επιθυμία υπάρχει. Ε, δεν είδαμε όμως ε, πολύ βιολετή χρώμα σε αυτά τα διαγράμματα τα οποία μας δείξατε και ο κύριος Χέτμαν μας είπε για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μεγαλύτερο το επίπεδο ε, στην Ισπανία, Γαλλία, ε, Ιταλία δεν έχουμε μεγάλη βελτίωση και η σύγκληση δεν είναι κάτι που πρέπει να λειτουργεί θεωρητικά, αλλά πρέπει να το βλέπουμε και στην πράξη η ευρωπαϊκή κρίση ε, θα ρίξω λίγο νερό στο μιλ του κυρίου Χαβι Λόπεφ τώρα ε, ξέρετε δεν έχουμε φύγει από την κρίση είμαστε ακόμα ε, στην κρίση και είπατε πολύ σωστά ότι αρκεί να αυξηθεί παραδείγματος χάρη τιμή του πετρελαίου για να βρεθούμε σε πολύ δυσχερή θέση. Επομένως ε, πρέπει να δούμε και ότι το ευρώ επιβαρύνεται ε, πάρα πολύ από όλα αυτά και υπάρχουν τελείως διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικές δομές ε, στην Ευρωζώνη και δεν θα πρέπει όλα αυτά να επηρεάσουν ε, το κοινό. Αυτό νόμισμα που ουσιαστικά περιορίζει και την πολιτική των κεντρικών τραπεζών, επιμικίνει και επιδεινώνει την κρίση. Επομένω, δεν θα πρέπει να αυταπατώμαθα ότι με τέτοια ε, ε, έγγραφα και με τη μεγαλύτερη σύγκληση θα λύσουμε όλα τα προβλήματα και θα καταθέσω και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρο για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους που συμβάλλανε στη συζήτηση αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για την απασχόληση στην Ευρωζώνη. Σήμερα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που κάνουμε ένα βήμα για την καταπόλεμηση της ανεργίας στην, στην Ευρώπη. Ας προσπαθήσουμε πραγματικά να το κάνουμε πιο δυναμικά, πιο ταραλέα και με αφοσίωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όχι μόνο για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όλοι δέχονται πια πώς η απασχόληση συμβάλλει στην ανάπτυξη των κρατών. Σε αυτή την Επιτροπή, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, κύριος Μοσκοβισή, μας είπε πως επιτρέπεται η παράκληση ακόμη και από τους πολύ σημαντικούς αυστηρούς κανόνες, το σύμφωνο σταθερότητα με την ρήτρα ευελεξίας, τις οποίες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ήδη κάνει η χρήση Ιταλία και η Ισπανία. Τι προβλέπει αυτή η ρήτρα. Δαπάνες που στοχεύουν στην απασχόληση να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ταπανών του σύμφωνο Σταθερότητας εάν έχουν θετικό εντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά του κράτους μέλος. Το ίδιο ακριβώς επισημαίνει και η Επίτροπος Απασχόληση κυρία Τάισεν απαντώντας σε ερώτηση 26 ευρωβουλευτών, πολλοί από τους οποίους είναι συνάδελφοι από αυτή εδώ επιτροπή και ρωτούσαμε την κυρία Τάισεν ακριβώς αν μπορούν να εξαιρούνται από το σύμφωνο σταθερότητας οι πόροι που κατανέμονται σε προγράμματα στήριξης ανεργίας. Η Επίτροπος απαντά επίσης και με κοινή συμφωνία ενός κράτους μέλος και της Επιτροπής μπορεί να υπάρχει ευελιξία όταν τίθεται σε εφαρμογή μίζωνος διαρτρωτικές μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Άρα, σας καλούμε να δούμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα αυτής της αλεπίδρασης, απασχόλησης και επίδρασης της στην, στις οικονομίας των κρατών μελών. Έκανα πρόταση μέσα της ομάδας μου GoNGL στους συντονιστές να ζητήσουμε σχετική έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και καθαρά μαθηματικό. Εγώ σε αυτήν την κατεύθυνση θα ήθελα να κινηθώ και να κάνω σχετικές προτάσεις στις οποίες εύχομαι και θα προσπαθήσω να δεχτεί ο εισηγητής και οι συνάδελφοί μου. Αλλά αφού έχουμε περάσει στη σφαίρα των μαθηματικών, επιτρέψτε μου να κλείσω μια μια του Αλβέρτου Αϊνστάιν. Ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος, όχι λόγω όσων κάνουν κακό, αλλά λόγω όσων παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ όχι απλώς να μην είμαστε μέρος της απραξίας, αλλά να μην είμαστε και συμμέτοχοι σε μια ανεπαρκή και υποκριτική μετριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους πρασίνους ή για το EFTD δεν βλέπω κανέναν, ούτε για το ΕΝΕ βλέπω κανέναν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Λουτσίντι θέλει το λόγο εκ μέρους της ε, Κομισιόν. Όχι. Έτσι κατάλαβα ότι δεν θέλετε το λόγο. Ωραία. Άρα, ο κύριος Λάγκεντέικ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τον κύριο Λόπε, την κυρία Τρεμπέσιου και την κυρία Κούνεβα. Για το σχέδιο έκθεση, τον και για τα σχόλια του υπολείπου. Και σίγουρα ε, καλό είναι να αντιμετωπίσουμε κοινού προκλήσει, να είμαστε πιο ανθεκτικοί, ανάπτυξη, ψηφιακέ δεξιότητε ε, κτλ. Ελπίζω ότι και εμεί από την πλευρά μα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε με βάση και συγκεκριμένες ενδείξεις ε, να σας δώσουμε δείκτες και να προβούμε στην αναγκαία έρευνα. Έτσι το βλέπουμε. Είναι κοινέ οι προκλήσεις. Κοινό κέντρο ερευνών, ένα θέμα συμπερίληψη κοινωνικού πυλώνα. Ευχαριστώ. Okay, merci. Donc, euh, en termes d'agenda, euh, la date τις διορίες για τις τροπολογίες. Λίγη στις 30 Αυγούστου. Οι τροπολογίες όμως πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά για να προλάβουμε. Το σχέδιο δράσης θα υποβληθεί, το σχέδιο έκθεσης του 24 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε 8 ή 9 Οκτωβρίου για να περάσει τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου η έκθεση του κ. Χέτμαν. Ευχαριστώ. Έχουμε προτρέξει κάπω, οπότε προλαβαίνουμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα μισή ώρα περίπου, γιατί στι 11 θα έρθει η κυρία Χάρτεκεν Κλάιν, τη Απασχόληση Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αυστρίας.

Υπότιτλοι Okay, and members. Αγαπητοί φίλοι και μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης και θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Χάρτιγκε Κλάιν, την Αυστριακή Υπουργό, που είναι Ομοσπονδιακή Υπουργό για την Απασχόληση, τις ε, κοινωνικές υποθέσεις, η υγεία και προστασία των καταναλωτών. Σχεδόν ε, ε συμπίπτει πλήρω το χαρτοφυλάκι όσες με τις δικές μας αρμοδιότητες. Μάλιστα, σε έχουμε ξανασυναντήσει. Ε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που σας έχουμε εδώ. Σας δίνω το λόγο λοιπόν για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας και το πρόγραμμα εργασιών σας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Χουλσκοκ, αξιότιμοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη τη Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, διερμηνείς από τις καμπίνες πίσω μου. Τους ευχαριστώ εκ των προτέρων για την διερμηνία. Χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι και μεγάλη τιμή που μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας ε, για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Αυστραϊκής Προεδρίας ε, στα θέματα τα κοινωνικά αναλαμβάνει η Αυστρία την Προεδρία στο τέλος αυτής της θητείας τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπω γνωρίζετε είναι μεγάλε οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φυσικά πολύ μεγάλε είναι και οι προσδοκίε και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Όλα αυτά ε, τα αντιλαμβανόμαστε. Γίνονται διαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή για το Brexit, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020 ε, και Έχουμε και ένα πολύ άλλο επίκαιρο ζήτημα, το ζήτημα της μετανάστευσης. Η κοινωνική ασφάλεια, η κοινωνική προστασία είναι ένας από τους πυλώνες, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του προγράμματός μας ε, για τον κοινωνικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ε, εκπροσωπεί ε, τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χρέος και λειτουργήμα. Ε, θέλουμε να εργαστούμε επικοδομητικά μαζί σας για το επόμενο εξάμεινο και αυτό πραγματικά είναι κάτι που το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα επί των οποίων υπάρχουν διαπραγματεύσει ε, ταυτόχρονα. Θα ήθελα να παραδείγματος χάρη να σας μιλήσω για την οδηγία για τις αποσπάσει των εργαζομένων. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ε, επίσης το θέμα των δίκαιων αποδοχών ε, και της ισότητας των συνθηκών εργασίας. Η τρίτη προεδρία ε, της Αυστριακής Παιδείας έχει ως σλόγγαν ε, «Η Ευρώπη που προστατεύει». Η Ευρώπη που προστατεύει αλλά και που είναι χρήσιμη ε, και σίγουρα οι δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους ε, και μια ευρύθμως λειτουργούσα αγορά, κινητικότητα, κοινωνική προστασία, υγεία, ασφάλεια στο χώρο εργασίας ε, και οι ελευθερίας μετακίνησης είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες. Υπάρχουν εργασιακά μοντέλα πρέπει να προστατεύσουμε, η ψηφιοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς πραγματικά Κινήσαμε τις εργασίες μας ε, με μεγάλη αφοσίωση και προσήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την Βουλγαρία και ιδίως ε, τον Υπουργό Πέτκοφ ε, για την εξαιρετική του εργασία. και όπως επιτάσσουν οι ε, αυστριακές παραδόσεις ε, θα εργαστούμε και εμείς, θα διαμεσολαβήσουμε ε, και θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε από κοινού το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προωθήσουμε το νομοθετικό έργο με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση ώστε τελικά ε, να σημειωθεί πρόοδος ε, και να ε, δώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη Προεδρία την Ρουμανία έχοντας επιτύχει στις προσπάθειές μας. Έχουμε διαπραγματεύσεις σε πολλά θέματα σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία και θέλουμε να κλείσουν όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με εσάς που είστε οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών, των ευρωπαϊκών πολιτών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ε, πρόοδο σε τρεις ε, σημαντικούς ε, τομείς, πρέπει να σου πω. Η Προεδρία μας θέλει να στηρίξει τη θέση του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του τριμήρους διαλόγου για τον κανονισμό 883 για την κοινωνική προστασία. Θέλουμε να υπάρχει συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων. Το Συμβούλιο τον Ιούνιο έδειξε συνεργάσιμο, έδειξε διάθεση συμβιβασμού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε μέτρα για την συμφιλίωση ε, της ε, επαγγελματικής ε, και προσωπικής ζωής και σίγουρα θα προωθήσουμε τις σχετικές διατάξεις. Το Συμβούλιο τον Ιούνιο επίσης ε, μετά από μικρής διάρκειας διαπραγματεύσεις κατάφερε να ε, οδηγηθεί σε μια κοινή θέση για μια οδηγία για διαφανείς ε, και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Έχουμε νέες μορφές εργασίας όπως είναι η εργασία σε πλατφόρμες ή η συμβάση μηδενικών ορών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη επισφάλεια και θέλουμε στο πλαίσιο των τερμερών διαλόγων να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι χρήσιμη, η οποία θα στηρίζεται ε, και θα προσφέρει μια ισορροπημένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε να προωθήσουμε την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Έχουμε αναλάβει δέσμευση να συνεχίσουμε τις ε, σχετικές διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου και να αντιμετωπίσουμε και τη μεγάλη πρόκληση της ψηφιοποίησης είναι αυτή η νομική πράξη κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφώνησαν επί του ε, κοινωνικού αυτού πυλώνα και δίνουν μεγάλη σημασία. Επίση, αλλαγέ ε, στι εργασιακέ διαδικασίε, δομέ απασχόληση, οργανώσει εργασία. Όλα αυτά οδηγούν ίσω και σε νέου κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων. Ο καρκίνο, ξέρετε ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εργασία. Θέλουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους, θέλουμε να περιορίσουμε την έκθεση. Αυτό είναι ένας σημαντικός στόχος που ξέρω ότι συμμερίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τη δεύτερη και την τρίτη δέσμη διαπραγματεύσεων για την οδηγία που αφορά τις καρκινογόνες ουσίες. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα για την Αυστριακή ε, Προεδρία. Θέλουμε λοιπόν γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε για τους εργαζομένους ε, επαρκή προστασία σε όλη την Ευρώπη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό για τις μεταλλεξιογόνες και καρκινογόνες ουσίες ε, με την Ολλανδία ε, έχουμε φτιάξει ε, τον οδικό χάρτη από το Άμστερνταμ στη Βιέννη και θα έχουμε μία συνεδρίαση στη Βιέννη για ε, το θέμα αυτό, για το θέμα του οδικού χάρτη από το Άμστερνταμ μέχρι την Βιέννη για τις καρκινογόνες όπως είπα. Επίσης, ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης, θα προωθήσουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Έχει ξεκινήσει σχετική προσπάθεια και θέλουμε να προωθήσουμε την προσθέμενη αξία μειώνοντα τι αλληλεπικαλύψει. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Αυστρία επίση είναι η ισότητα και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα για τα άτομα με αναπηρία, να μειώσουμε τους φραγμούς ε, ε, και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις όπλες του τριμερούς διαλόγου που ξεκίνησαν επί Βουλγαρικής Προεδρίας για να κλείσουμε ελπίζοντας αυτό το φάκελο και θα υπάρξει και μια συνεδρίαση, μια ημερίδα των συνηγόρων του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με θέματα αναπηρίας στην Ευρώπη. Επίσης, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, έχουμε προγράμματα τομεακά, τα οποία θέλουμε να τα σχετίσουμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και έχουμε και τις στάσεις αναχώρα, την αρχή, ε, μάλλον ε, τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Με όλα αυτά έχει ξεκινήσει ένα νέο μονοπάτι, το οποίο χάραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε και το νέο πρόγραμμα για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο σχηματισμό του Συμβουλίου, το οποίο θα προεδρεύω. Επίση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με τι ε, διαπραγματεύσεις ε, του Ιούλιο θα ξεκινήσουμε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα κοινωνικά ζητήματα και θέλουμε να παραμείνει ε, το Ταμείο αυτό ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο τώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, θα ε, συνεχίσουμε με το πακέτο του φθινοπόρου το Δεκέμβριο να ασχολούμαστε ε, με τα θέματα που άπτονται της απασχόλησης και συγκεκριμένα έχουμε την ετήσια επισκόπηση για την απασχόληση και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσουμε και να επεξεργαστούμε. Επίσης, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα ζητήματα του κανονισμού που αφορούν τους οργανισμούς όσα Eurofound και Σεντεφόπ. Θέλουμε να κλείσουν οι σχετικές ε, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο τριμερούς ε, διαλόγου. Τώρα, θέλω να πω ότι θέλουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα της Τρόικας ό,τι αφορά την άτυπα απασχόληση και να θα εστιάσουμε στα κοινωνικά ζητήματα, θα εστιάσουμε στην εργασία, θα εστιάσουμε στην ψηφιοποίηση, ε, στην ελάφρυνση ε, και σε κάποιες ε, βελτιώσεις των συνθήκων εργασίας, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, κοινωνική προστασία, που καθακαλύπτει και τις νέες μορφές απασχόλησης ποιότητα εργασίας. Υπάρχει, ε, υπάρχει μια άτυπη συνεδρία των Υπουργών Απασχόλησης Κοινωνικής Πολιτικής 19 και 20 Ιλίου στη Βιέννη. Εκεί θα δούμε την ατυπική εργασία. Ε, πάντοτε έχοντας υπόψη μας τα θέματα της ψηφιοποίησης ε, και των πλατφορμών ε, που είναι μια νέα εξέλιξη στον χώρο της εργασίας. Και αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι ε, η κοινωνική προστασία, το δικαίωμα των ανθρώπων στην εργασία. Πρέπει όλα αυτά ε, να καλύπτονται με αναλογικό τρόπο στο πλαίσιο των νέων μορφών εργασίας. Θέλουμε να προωθήσουμε και να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές, τα καλά παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, αυτοματισμός, τα ρομπότ που μπορούν να βελτιώσουν τις, και να αλλάξουν άρδιν τις συνθήκες εργασίας και την καθημερινή εργασία. Επίσης, στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, ε, τα πλεονεκτήματα θα τα συζητήσουμε, αλλά και τους κινδύνους και ε, θα παρουσιάσουμε μία έκθεση που θα δίνει παραδείγματα των νέων τεχνολογιών ε, και θα σας καλωσορίσω με μεγάλη χαρά ε, στις διάφορες αυτές συνεδριάσεις που οργανώνουμε. 19 Σεπτεμβρίου έχουμε μια υψηλού επίπεδου συνεδρίαση με θέμα την ψηφιοποίηση και το απασχόληση 4.0 και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωβουλευτές. Αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ε, ε, πραγματικά έχουμε σημαντικές προκλήσεις ε, και έχουμε πολύ κοινή δουλειά να κάνουμε στο δεύτερο εξάμεινο του 2018. Προσβλέπω στη συνεργασία μας. Ε, πιστεύω θα είναι στενή, θα είναι καλή συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Minister. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και Κλάιν. Περνάμε στους συντονιστές τώρα ή στους αντικαταστάτες τους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Χάινς Μπέγκερ, που είναι Αυστριακός και μέλος του, της Επιτροπής Απασχόλησης και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την, ε, που μου δίνετε το λόγο, ε, επειδή είμαι και ε, της ίδιας επικότητας με την ε, πρόεδρο την Προεδρεύσα του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε σε σχέση με την Αυστριακή Προεδρία που συνοδεύεται από πολύ μεγάλες ε, προσδοκίες ε, γιατί είναι η τελευταία ολοκληρωμένη Προεδρία πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές που είναι το Μάιο του χρόνου και σας μας είπατε ποιο είναι το σλόγγαν σας, μια Ευρώπη που προστατεύει και σίγουρα αυτός είναι ο απότατος, ο ύψιστος ε, στόχος και Φυσικά κοινωνική προστασία εντάσσεται σε αυτή την προστασία τη γενικότερη που θέλουμε να παρέχει η Ευρώπη. Είπατε και εσείς ε, ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Σίγουρα ε, οι εργαζόμενοι με αναπηρία ε, εστιάζεται σε αυτούς τους εργαζομένους και αυτό το χαιρετίζω ιδιαίτερα. Υπάρχουν τεράστιες ψηφιακές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η Αυστριακή Προεδρία επίσης είναι καλό που δίνει προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν κίνδυνοι αλλά κυρίως ευκαιρίες για την ποιότητα, ε, για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων. Είναι πολύ θετικά τα όσα θα μπορούσαν να προκύψουν. Ε, είναι σημαντικά όλα αυτά και συμφωνώ με τις προτεραιότητες αυτές της Αυστριακής Προεδρίας. Ένα άλλο επίκαιρο, ε, πολύ επίκαιρο ζητήμα που μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή μας πολύ συχνά είναι οι, βιώσιμες, ε, συγγνώμη, διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας ε, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, για την κοινωνία. Και το ερώτημά μου είναι η Αυστριακή Προεδρία. τι άποψη έχεις ότι αφορά την προστασία των εργαζομένων που εργάζονται σε επισφαλείς, με επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο αυτών των συνθήκων, των προβλέψεων και των διαφανών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους υπόλοιπους συντονιστές, ε, παρακαλώντας τους να μην υπερβούν το δίλεπτο. Η κυρία Χογγέριου από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Θα βάλω τα δυνατά μου, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είχαμε ήδη συναντηθεί στη Βιέννη, παρασκευάζοντας αυτή τη συνάντηση. Ε, διάβασα το πρόγραμμα της Αυστηριακής Προεδρίας γιατί σκέφτηκα, σήριξω μια ματιά για να δω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Αυστρίας. Και όταν διάβασα το πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας, διαπίστωσα ότι πολλά από τα τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών σας και πραγματικά ελπίζω να καταφέρετε να φέρετε σε αίσιο πέρα όλα αυτά τα ζητήματα. Με εξέπληξε κάπως ε, που παρελείπεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Χαίρομαι όμως που το αναφέρατε στην ομιλία σας. Γιατί νομίζω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να έχω, εξασφαλίσουμε συνθήκες θεμητού ισότιμου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόμενους. Φαίνεται ότι παρεξήγησα την παράληψη της Ευρωπαϊκής Αρχής εργασίας σας, ε, της ευρωπαϊκής εργασίας ε, από το πρόγραμμα εργασιών σας. Το ερμήνευσα ως αδιαφορία της Αυστρικής Προεδρίας, αλλά με διαψεύσατε. Είπατε ότι σας ενδιαφέρει το θέμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και ελπίζω με το που θα ολοκληρωθεί η Προεδρία να ε, σταθεί να συστηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και να γίνει και λειτουργική αμέσως. Όπω είπε ο κύριο ε, Μπέκερ, μα ενδιαφέρουν διαφανεί και προβλέψιμες εργασιακέ συνθήκε για όλους τους εργαζόμενους. Στη σχετική οδηγία, το Συμβούλιο τον Ιούνιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση που αποκλείει όμως τους πιο ευάλωτους ε, εργαζόμενους. Αυτούς που δουλεύουν ε, με συμβάσεις ελάχιστων ή μηδενικών ωρών γιατί το Συμβούλιο απέκλεισε αυτές τις συμβάσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εμείς προτείναμε μια ευρωπαϊκή απαγόρευση, ολοσχερή απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών ορών. Εσείς τι γνώμη έχετε. Είστε πρόθυμοι και πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να στρέψετε τον τριμερή διάλογο προς σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κυρία Μάκιντάιρ από τους ε, συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την Υπουργό στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Ε, Εξετάζοντα τι προτεραιότητε τη Αυστριακή Προεδρία, διαπιστώνουμε ότι έχετε ένα μακροσκελή κατάλογο σημαντικών προτεραιοτήτων που απηχούν και τις δικές μας προτεραιότητες, ε, ισορροπία ιδιωτικής επαγγελματική ζωής, προστασία από καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες ουσίες, προσβασιμότητα, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες. Οπότε έχω δύο ερωτήσεις. Μας ενδιαφέρει μια σωστή νομοθεσία που θα είναι εφαρμόσιμη και εφικτή. Έχει νόημα λοιπόν να προωθούμε ταυτόχρονα τόσε πολλέ φιλόδοξε νομοθετικέ προτάσει, ενώ πλησιάζουμε προ την λήξη των αντίστοιχων θητιών μας. Προβληματίζομαι και παρά τις αγαθές μας προθέσεις να προωθήσουμε ε, νομοθετικές προτάσεις πάση θυσία μόνο και μόνο χάρη συμφωνίες πριν ολοκληρώσουμε την κοινοβουλευτική μας θητεία. Είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Μήπως καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθούμε ε, σε λίγα και καλά αλλά σε πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές ε, συζητήσεις. Ό,τι αφορά τον κοινωνικό πυλώνα δικαιωμάτων, οδήγησε σε πολλέ νομοθετικέ προτάσει που επεξεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία και την ε, προτινόμενη οδηγία για διαφανεί και προβλέψιμε εργασιακέ συνθήκε. Δεδομένου όμω ότι πρόκειται μόνο για πολιτική διακήρυξη προ το παρόν, ε, φαίνεται ότι έχει λάβει και άλλε διαστάσει με αυτέ τι νομοθετικέ προτάσει. Και αν δούμε πόσο συχνή μνήμα των δικαιωμάτων γίνεται στι πρόσφατε νομοθετικέ προτάσει. Ε, υπενισόμαστε το δεσμευτικό χαρακτήρα ουσιαστικά του κοινωνικού πυλώνα. Και ε, κατοχυρώνουμε τέτοια δικαιώματα και αντίστοιχε υποχρεώσει. ενώ κανονικά ο κοινωνικό πυλώνας έχει απλώς διακηρυκτικό χαρακτήρα. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλβέ Σαμπόν από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την ε, Υπουργό που ήρθε να μας μιλήσει και να μας ακούσει και ευχαριστώ για την ενέργεια που έχετε επιδείξει μέχρι στιγμής και τον ενθουσιασμό σα. Λίγα λεπτά έχω γι' αυτό θα επικεντρωθώ στα ουσιώδη. Δεν προλαβαίνουμε για να αναφερθούμε λεπτομεριακά σε κάποια θέματα. Πάντως το χαρτοφυλάκιό σα ε, θα έχει τεράστια σημασία στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για το υπόλοιπο τμήμα της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Για δύο κυρίως λόγους. Γιατί αναλαμβάνετε την Προεδρία τη στιγμή που το κοινωνικό θεματολόγιο, όπως είπε η κυρία Μακεντάιρ, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και ποσοτικά. Γιατί η κοινωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν ο κοινωνικός πυλώνας ή ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που αποφασίστηκαν στο Γκέτεμπορκ να μετατραπούν, να λάβουν σάρκα και ωστά σε συγκεκριμένα μέτρα που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό και τα κοινωνικά ζητήματα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Στο παρελθόν ήταν τα οικονομικά που είχαν τα πρώτα. Τώρα τα κοινωνικά ζητήματα αναδείχθηκαν περισσότερο. Γι' αυτό και ο ρόλο σα θα είναι θεμελιώδη και κρίσιμο επίση. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Γι' αυτό και το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο και ενδιαφέρει του πάντε. Γιατί όλοι προσβλέπουμε σε αυτά αποτελέσματα που θέλουμε να παρουσιάσουμε στου Ευρωπαίου πολίτε για τα ζητήματα που του προβληματίζουν. Την απασχόληση δηλαδή και τα κοινωνικά θέματα. Αυτό θα πρέπει να το έχετε κατά νου. Γιατί πραγματικά όλοι επιθυμούμε κάποια σκέρις νομοθετικές προτάσεις να διεκπαιρεωθούν στη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική θητεία, πριν αναλάβει το επόμενο κοινοβούλιο. Γι' αυτό και θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια επιλογή, μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Εγώ είμαι ο συντονιστής ε, για τα θέματα προβλεψιμότητα ε, των εργασιακών συνθήκων και διαφάνεια. και είμαι και εισηγητή για τους οργανισμούς ε, Eurofound και ούτω καθεξή. Βέβαια δεν έχουν όλα τη ίδια σημασία. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία, στι εργασιακές συνθήκε, στο συντονισμό τη κοινωνική ασφάλεια και στην εξισορρόπηση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, πραγματικά θα μας ευχαριστήσουν οι πολίτες. Σας ευχαριστώ κύριε Καλβέσομπο. Για την κούε κάποιος. Όχι. Από τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή Απασχόληση. Χθε είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον συνάδελφό σας ε, κύριο Στράου ε, και στην Περιφερειακή Επιτροπή και στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Δύο σημαντικέ επιτροπέ για τα κοινωνικά δικαιώματα για την κοινωνική Ευρώπη. Η οικοδόμηση τη ε, κοινωνική Ευρώπη, η ενίσχυση τη κοινωνική Ευρώπη είναι πιστεύω κάτι που θέλουμε όλοι να προωθήσουμε. Είπατε Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό είναι το σλόγγαν και πραγματικά περιέχει πολλά αυτό το σλόγγαν, όπως πολλά περιέχει και το πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας και για το θέμα της απασχόλησης ε, είχα κάποια απογοήτευση και εγώ νιώσει διαβάζοντας το πρόγραμμα, αλλά εσείς μας ε, καθυσυχάσατε σήμερα στην παρουσίασή σας. Επίσης, αυτή η Ευρώπη ε, προστατεύει, αλλά υπάρχει και το θέμα της μετανάστευσης, προστασία εξωτερικών συνόρων που είναι στο προσκήνιο και η κοινωνική προστασία, η προστασία των εργαζομένων, η προστασία του κλίματος, οι οικολογικέ θέσει εργασία, η δημιουργία θέσεων εργασία είναι σημαντικά θέματα, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ ε, μπει στην πρώτη γραμμή, έχουν επισκιαστεί από τα ζητήματα που προανέφερα, μετανάστε κτλ. Εσεί θα αλλάξετε αυτή την κατάσταση, δηλαδή θα βάλετε στην πρώτη γραμμή την κοινωνική Ευρώπη, την κοινωνική προστασία, γιατί μιλήσατε επίση όχι για μόνο για μια Ευρώπη που προστατεύει, αλλά και που είναι χρήσιμη. Χρήσιμη για του πολίτε, ε, για άντρε, γυναίκε, για εργαζομένου. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση το ρόλο ε, ε, της ε, ουδέτερης Αυστρίας που είπατε ότι οικοδομείται συνεργασία. Αυτός είναι ο ρόλος της Αυστρίας να είναι ένας διαμεσολαβητής, ένας ουδέτερος διαμεσολαβητής. Πώς τον αντιλαμβάνεστε αυτό το ρόλο. Ε, διότι ε, υπάρχει ε, μια μαζική επίθεση σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, το θέμα της, του κατοίκων εργασίας, όλα αυτά παίρνουν μια ευρωπαϊκή διάσταση και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα με τον ε, ε, Υπουργό στην Αυστρία έχουμε ανησυχίες και τι γίνεται με τα οικογενειακά επιδόματα, τι γίνεται με την απασχόληση των ε, γυναικών που είναι και μητέρες. Εσείς ναι μεν θέλετε να έχετε μια ουδέτερη θέση, να θέση να ουδέτερο διαμεσολαβητή, αλλά ε, νομίζω ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, συνολικά εσείς θα είστε αυτός ο διαμεσολαβητής ουδέτερος που είπατε, αλλά δεν ξέρω αν η υπόλοιπη κυβέρνηση θα μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Επίσης για τους πρασίνους ε, μας ενδιαφέρει να έχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, ε, τη συμμετοχή των τοπικών περιφερειακών φορέων στο πλαίσιο της ε, αρχής της εταιρική σχέσης και στον προγραμματισμό. Πώς λοιπόν θέλετε να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών, κοινωνική εταίρη, τοπική περιφερειακή φορείς, στη διαμόρφωση αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ και τι χρονοδιάγραμμα έχετε προβλέψει. Τελευταία ερώτηση. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την κοινωνική πολιτική για το επόμενο εξάμεινο και την Αυστριακή Προεδρία είναι το πολιτής πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερο λυπηρό το ότι ο συνάδελφό σα, ο Υπουργό Λέγκερ, δεν έρχεται αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Προπολογισμών. Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε πολλές επιτροπές και ο Υπουργός ε, Λουγκίν δεν έρχεται στην πολύ σημαντική Επιτροπή Προπολογισμού για το πολύ σημαντικό θέμα ε, του προϋπολογισμού ε, και έχουμε τις διαπραγματεύσεις του πολιτές μεσονομικό πλαίσιο με σημαντικό στοιχείο το θέμα της πολιτικής συνοχής που απειλείται με μείωση των κονδυλίων κατά 45% ε, και έχουμε κάποιες ε, χώρες ε, που θίγονται, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού στον τομέα άμυνας και προστασίας των συνόρων. Αυτή η τρομερή μετατόπιση των κονδυλίων από την κοινωνική συνοχή στην πολιτική άμυνας Θεωρείτε ότι είναι κάτι λογικό. Δεν θα πρέπει να μπουν κονδύλια για την υποστήριξη της κοινωνικής Ευρώπης. Η FDD δεν εκπροσωπείται σήμερα. Οπότε πηγαίνουμε στον κύριο Ντομινίκ Μαχτά από το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίζω και τη νέα Αυστριακή Προεδρία. Είμαι θα ιδιαίτερα ευτυχής εδώ που μας παρουσιάζετε τις προτεραιότητές σας. Θα είμαι σύντομος, θα σας θέσω δύο ερωτήσεις. Από την 1η Ιουλίου, εδώ και δέκα μέρες δηλαδή, μετά από ένα δημοψήφισμα του 2014, η Ελβετία επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στις ε, οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τις κενές θέσεις από Ελβετούς πολίτες. Θέλετε να κάνετε το ίδιο στην Αυστρία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συλλέγει πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για τον ετήσιο αριθμό των θέσεων απασχόλησης που δίδονται στους Ευρωπαίους πολίτες ανέργους και που στο παρελθόν τις θέσεις αυτές τις κατήχαν πολίτες ε, μη κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση για τον έλεγχο των συνόρων. Μάθαμε ότι στην Γερμανία μόνο το 10 με 15% των μεταναστών που έφτασαν το 15 κάτω από 13% full time ενώ η Γερμανία έχει ξοδέψει 15 δις για να τους υποδεχτεί. Στην Γαλλία εμείς αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές τρομερές τρομοκρατικές ενέργειες. Για τα δύο αυτά προβλήματα πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στα σύνορα τα εσωτερικά των κρατών μελών όπως στη δική σας χώρα προς ποια επιλογή θα κατευθύνεται τις εργασίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Έχετε πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις, έχετε δεχθεί πολλές και υπάρχουν άλλα εννέα μέλη που θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Και γι' αυτό παρακαλώ εάν είναι δυνατόν να είσαστε πάρα πολύ ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ευχαριστώ. Θερμά θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Κάποιοι έβαλαν πολύ άριθμα ερωτήματα και αν ξεχάσω κάποια ερωτήματα προκαταβολικά συγγνώμη. Θα προσπαθήσω όμως να τα απαντήσω όλα. Και ξεκινώ με τον βουλευτή Μπέκερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας εισαγωγικά λόγια, αλλά και για τις ερωτήσεις που μου θέσατε για την προστασία των επισφαλών ε, εργαζομένων. Σίγουρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε την πρόταση ε, για τις νέες μορφές εργασίας που πρέπει να καλύπτονται ε, και οι συμβάσεις ε, μηδενικών ορών περιλαμβάνονται σε αυτές τις νέες μορφές. Δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Αυστρία. Εμείς θέλουμε επίσης με την ψηφιοποίηση ε, να προχωρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το Σεπτέμβριο οργανώνουμε, όπως είπα, ίσως το ανέφερα νομίζω, θα έχουμε ένα συνέδριο για τα θέματα της ε, ψηφιοποίησης. Το δεύτερο για την κυρία Γιονγκέριους, ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης. Αξιότιμη κυρία Γιουγκέριους, ε, είμαστε όπως γνωρίζετε στην αρχή της διαδικασίας και υπάρχουν ακόμη ανοιχτά πολλά ερωτήματα. Στόχος της Αυστριακής Προεδρίας ε, είναι ε, να ε, σημειωθεί σημαντική πρόοδο στο θέμα της ίδρυσης αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης. Ε, επίσης, το θέμα των κρατών μελών θα, τα, ασχοληθούμε με όλα αυτά και σίγουρα θέλουμε να υπάρχει μια καλύτερη ροή πληροφοριών για τα διοσυνεριακά ζητήματα και για την το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να σημειωθεί πρόοδος. Για την κυρία Μάκιντάρ, συγγνώμη, δεν έχω συνηθίσει κάποια ονόματα. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι μας ενδιαφέρει πιο πολύ ποιότητα ε, από ότι η ποσότητα. Σίγουρα είναι όμως μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτων ευρωεκλογών και καλό είναι να καταφέρουμε να κλείσουμε στο δυνατόν περισσότερα ανοιχτά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η Ευστρική Προεδρία θέλει ε, να προωθήσει ε, τα θέματα που άπτονται των κοινωνικών δικαιωμάτων, ε, να έχουμε τις προβλέψιμες και διαφανείς συνθήκες εργασίας, την αρχή της απασχόλησης, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία ε, για τους εργαζομένους. Όλα αυτά θα τα επεξεργαστώ, με, όπως είπα, με τις καλύτερες των προθέσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε και θα εξετάσουμε, όπως είπα, και την ετήσια επισκόψη για την απασχόληση μέχρι το Δεκέμβριο. για να προωθήσουμε ακριβώς αυτό τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σίγουρα είναι στο επίκεντρο ε, οι διαπραγματεύσει ε, για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για μας ε, προτεραιότητα είναι το ΕΚΤ-ΣΥΝ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΣΥΝ, αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε να έχει επίσης επαρκή κονδύλια η πολιτική απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων και όλοι μαζί θα εργαστούμε για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμπόν. Και εδώ επαναλαμβάνω ποιότητα, ποσότητα, φυσικά για μας έχει προτεραιότητα ή ποιότητα, όμως ε, θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν ε, περισσότερα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών. Ε, έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητές μας, σίγουρα ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, το είπα από την αρχή, είναι μία από τις προτεραιότητες. Για την κυρία Βάνα που έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες ό,τι αφορά το πρόγραμμα Αυστριακής Προεδρίας. Ε, περιλαμβάνει ε, όλα τα σημεία τα οποία ε, είναι στο χαρτοφυλάκιό μας. Η κοινωνική Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως η συμφιλίωση και επαγγελματική προσωπικής ζωής, ψηφιοποίηση και σχετικές προκλήσεις. Ε, τώρα για τα εθνικά ζητήματα, στα οποία αναφερθήκατε, θα μου τρέψετε να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είμαι μια ουδέτερη διαμεσολαβήτρια, όπως είπα, και το ίδιο ε, ισχύει ε, και εδώ δεν θα μιλήσω καθόλου για εθνικά ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, από αυτό το βήμα. Επίσης, ε, το ότι ε, είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση για να παραμείνει κανεί ένα πραγματικά έντιμο και ουδέτερο διαμεσολαβητή. Θα προσπαθήσω να έρθω στο ύψο αυτή τη πρόκληση. Επίση, ό,τι αφορά ε, οικονομικές πτυχές ε, ε, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες ε, για το πολιτές μεσομικό. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα που θα πρέπει να αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όπως είναι η κατανομή, τα ποσά και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα παρακολουθούμε από κοντά τα θέματα που άπτονται του δικού μας χαρτοφυλακίου. Φυσικά ε, θα ενημερώνουμε τους ευρωβουλευτές ε, για οποιαδήποτε πορίσματα και αποτελέσματα των ε, διαφόρων σχηματισμών του Συμβουλίου και φυσικά και ο Πρόεδρος Ταγιάννη έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή πάντοτε στο πλαίσιο αυτών των Συμβουλίων με τους αρχηγούς κρατών και κυβέρνηση για τους μεταφέρει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και σίγουρα θα έχουμε υπόψη σε όλα αυτά που είπατε για ε, την εφαρμογή του προγραμματός μας. Ό,τι αφορά το εκτ ε, και τη διαμόρφωση αυτού του νέου ταμείου στο πλαίσιο των διαθροτικών τομείων, σίγουρα ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις και απαιτήσει για τον τομέα της πολιτικής απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής. Θα συνεργαστούμε και με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Βιωσιμότητας. Επίση, έχουμε άτυπη συνάντηση τον Ιούλιο για τη ψηφιοποίηση. Θα συζητήσουμε εκεί όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και το έκτε ΣΥΝΑ. Και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο επίσης θα έχουμε ε, άλλη ενημέρωση. Πάντως ε, πρέπει να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Τον κύριο Μαχτρά θέσεις εργασίας ε, στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το βασικό θέμα της παρέμβασής σας. Σίγουρα ε, και οι βασικές ελευθερίες ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες, ελευθερία κυκλοφορίας, ιδίως των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, σίγουρα το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους Έχουμε την μπλε κάρτα επίσης ε, που ρυθμίζει ε, ε, τις διαδικασίες. Τη Δευτέρα θα τα συστήσουμε με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Κίκλ. Ένα άλλο ερώτημα ήταν η ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Οι διαβουλεύσεις ε, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ε, ασύλου θα συνεχιστούν και επί Αυστριακής Προεδρίας. Τη Δευτέρα θα τα δω, όπως σας είπαμε, τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Κίκλ. Σίγουρα υπάρχει το θέμα της ζήτησης εργατικού δυναμικού και εδώ ε, είναι ένα θέμα που συνδυάζεται και συνδέεται με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό γιατί υπάρχει πράγματι ανάγκη για εξειδικευμένο εργατικό ε, δυναμικό. Θέλουμε ε, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, απασχόληση των περισσότερων <clears throat> μεταναστών και προσφύγων για να ελαφρύνουμε και τα κοινωνικά συστήματα, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστώ. Thank you, Klein. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον επόμενο κατάλογο τώρα των ερωτήσεων. Η συμπατριώτη σας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, τα σημαντικά ζητήματα ε, είναι αντικείμενο ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, τα λιγότερο σημαντικά εθνική διαπραγμάτευση. Η απασχόληση, η ασφάλεια, η προστασία των θέσεων εργασία, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για του ε, Ευρωπαίου πολίτε. Μέχρι στιγμή ε, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο του, της απασχόλησης, ε, είχαμε ε, και στην προηγούμενη Αυστριακή Προεδρία ε, πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή επίδοση. Έχω κάποια ερωτήματα, καταρχάς σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Αγοράς Εργασίας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι δεσμευτικό. Εσείς είχατε πει στο Αυστριακό Κοινοβούλιο ότι αυτή η Ευρωπαϊκή ε, Αρχή ε, θα σημαίνει μερισσότερη γραφειοκρατία και δεν θα προσφέρει προστιθέμενη αξία. Τι από τα δύο τελικά γιατί στην λίστα προτεραιότητας του προγράμματος ε, της Αυστριακής Προεδρίας ε, δεν το βλέπουμε. Ποια είναι η θέση σας τελικά. Είναι ε, ένα hot spot ε, για κοινωνικό dumping και εργασιακό dumping. Ε, η Αυστρία δεν θα ήθελα να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσουμε για τα θέματα work-life balance, ισορροπία επαγγελματική προσωπική ζωή. Τι άλλο καλύτερο από αυτό. Είναι ένα θέμα που προστατεύει και φροντίζει και είναι χρήσιμο για, την, για τους πολίτες. Πώς θα προχωρήσουμε. Λέτε πιο πολύ ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τα ρυθμίσουν αυτά. Εδώ όμως θέλουμε να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή διάσταση. Υπάρχει προσθέμενη αξία και μπορούμε ε, να προβάλλουμε αυτή την ευρωπαϊκή αξία στους Και το τρίτο θέμα, το gold plating, ο κανονιστικός υπερθεματισμός. αυτά τα οποία εμεί υποστηρίζουμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, δεν έχουν κάνει τίποτα με το τι γίνεται στην Αυστρία που έχουμε 12 ώρο ε, την εβδομάδα, 60 ώρο την εβδομάδα στην Αυστρία και ε, ουσιαστικά κατάλυση πολλών κοινωνικών ε, δομών και δικαιωμάτων. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Ε, θέλουμε να κατοχυρώσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, να έχουμε καλύτερα πρότυπα. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα συνονθήλευμα, ένα αμάγλγαμα. Πώς θα τα δείτε όλα αυτά, αποφεύγοντας και τον κανονιστικό υπερθεματισμό. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και για την προθυμία σας να απαντήσετε. Επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, γιατί είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα στην Ευρώπη είναι να μπορεί κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει μια αξιοπρεπή θέση εργασίας. Και αυτή είναι ε, η θεμελιώδης πρόκληση όχι μόνο της κοινωνικής ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Και σίγουρα ο κοινωνικός πυλώνας ε, μιλάει για την κοινωνική προστασία, τις ε, δικαιότερες εργασιακές συνθήκες, και αυτές οι προκλήσεις που είναι ουσιαστικά τρεις σε μία είναι η πιο κρίσιμη αποστολή της Προεδρίας. Ναι, παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο. Και επίσης περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να συμπληρώνει τις, Ευρωπαϊ... τις Εθνικές Αρχές Εργασίας, δηλαδή να προωθεί πληροφορίες και καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν δραστικές διακρίσεις, εκμετάλλευση, κοινωνικές απάτες, πολλές και διάφορες μορφές ε, καταστρατήγησης όχι μόνο στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Στη Βιέννα ε, έχει την έδρα του ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, φρά και έχει καταδείξει κατάφορη παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας και εκμετάλλευση των Ευρωπαίων εργαζομένων. Οπότε θα ήθελα η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, να κατοχυρωθεί, γιατί είναι πραγματικά η κατάλληλη αρχή ε, για να καταστήσει αυτή την ε, εθελοντική κινητικότητα των εργαζομένων συναφή με τις αξιοπρεπείς και δίκες εργασιακές συνθήκες. Επίσης, ό,τι αφορά την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ε, επιδομάτων των οικογενειακών για τα παιδιά. Η αυστρική κυβέρνηση ε, επιμένει να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το συμπεριέλαβε στην ε, αρχική της πρόταση για τη συντονισμό σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας. Και παρόλο που και η Βουλγαρική Προεδρία δεν συμπεριλάβε το θέμα αυτό στα μερικά συμπεράσματα που συμφώνησε. Είπατε ότι οι τοπικές και εθνικές πολιτικές δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την Αυστριακή Προεδρία και το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι αυτό το θέμα τελικά δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασιών της Αυστριακής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Μαρία Ντουιάννα. me réjouis euh, Βλέπω ότι η θεματολογία αυτή ανήκει στις προτεραιότητές σας. Στη Βουλγαρική Προεδρία την τελευταία στιγμή δόθηκε μια εντολή διαπραγμάτευσης. Ελπίζω ότι για τον τριμερή διάλογο η εντολή αυτή να οδηγήσει σε μια λύση η οποία έτσι και αλλιώς προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια πρωτοβουλία για την συμφιλίωση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει ότι η διαβούλευση αυτή δεν θα πρέπει να ενισχύσει τα παραδοσιακά πρότυπα τα οποία εγκλείουν την γυναίκα σε ένα αυστηρά οικογενειακό ρόλο κάτι το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω διακρίσει στον τομέα της απασχόλησης, το μισθολογικό και τον συνταξιοδοτικό. Συνεπώς λοιπόν ο συνδυασμός αυτός πρέπει να ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Σημερίζεστε την πρόταση την οποία έχει, κάνει, έχει προτείνει για συζήτηση η Μαρία Τάισεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι μόνο ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, αλλά και έλλειψη διακρίσεων εις βάρος των γυναικών γιατί η γονική άδεια ε, λαμβάνεται κατά 87% από τις γυναίκες και όχι από τους άνδρες σήμερα. Λοιπόν, δεν ε, ζητώ την γνώμη της χώρας σας, αλλά ως Προέδρου ε, είστε υπέρ του ελαχίστου παρανομαστού, κοινού παρανομαστού ευρωπαϊκού προτύπου έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον συνδυασμό της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής. Αν θέλαμε εμείς να διαλέξουμε ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένειά μας, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην οφείλουν να αποφασίσουν ανάμεσα στη δουλειά και στην οικογένεια. Ευχαριστώ Κόζα. Πρόεδρε, ευχαριστώ επίσης και την ε, κυρία Υπουργό. Θα θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, σύντομα, ο βούλγαρος συνάδελφος ήδη αναφέρθηκε για την συνεργασία και τον συντονισμό σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση και σε σχέση με τις δυνατότητες κοινωνικής ασφάλισης και των υπολείπων μελών της οικογένειας. η Αυστρία ως χώρα μέλος πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες οι οποίοι εργάζονται στην Αυστρία, τον οποίων όμως τα μέλη των οικογενειών τους ζουν σε μια άλλη χώρα μέλος. Πώς μπορούν λοιπόν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να λαμβάνουν τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι το συμβατό με τις νομοθετικές μας πράξεις και με το κοινοτικό κεκτημένο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς θα μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα αυτό. Έχετε κάποιες απόψεις σαν Αυστρία, χώρα μέλος, αλλά αυτό δεν επιτρέπει ας πούμε την τιμαριθμοποίηση των συγκεκριμένων επιδομάτων. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία. Ο πέμπτος τριμερής διάλογος έγινε χθες και βασικό θέμα για συζήτηση ήταν ε, η νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα. Χαίρομαι που άκουσα από πλευρά σας ότι είναι μια σημαντική προτεραιότητα και ότι επιθυμείτε να κλείσει το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατόν, αν και μένουν ορισμένα χαίνοντα σημαντικά θέματα. Δεν θα περάσω τώρα στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω ε, με ποιο τρόπο εσείς αντιμετωπίζετε την πράξη αυτή για την προσβασιμότητα. Υπάρχουν 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που περιμένουν την πράξη αυτή που καθυστερεί εδώ και 10 χρόνια. Σομπόρ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σχετικά τώρα με τα επιδόματα, τα οικογενειακά και την τιμαριθμοποίησή τους και εγώ θα ήθελα να θέσω το ίδιο ερώτημα προς τους συναδέλφους. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί πολίτες επίσης οι οποίοι εργάζονται φροντίζοντας τους ηλικιωμένους στην Αυστρία που δεν είναι Αυστριακοί. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν τους ίδιους φόρους για τις αμοιβέ τους και σχετικά λοιπόν με τα οικογενειακά επιδόματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον χώρο, την χώρα στην οποία ζει, το, ζουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους. Η κυρία Κοζόφσκα Ραγεύητς παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την Υπουργό για την παρουσία της εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ τι θα γίνει με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών επιδομάτων. Γιατί εμεί στείλαμε επιστολή μαζί με άλλε συναδέλφου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική ερώτηση και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη ότι ε, είναι πολύ επιμαχό το θέμα και δεν θα συμπεριληφθεί και η ίδια ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προκαλέσει έντονε διαμαρτυρίε. Η Αυστριακή Προεδρία πόσο σκοπεύει να επιλύσει αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και τι λύση θα προτείνει. Δεύτερη ερώτηση για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Εδώ έχουμε ένα τυχό θέμα. Ε, είναι ε, μεγάλη υποεκπροσώπηση των ε, γυναικών στην αγορά εργασία ανάλογα με τις προσδοκίες τους, ε, τη μόρφωσή του, Έχουμε κενό 11% και 17% μισθολογική διαφορά, διαφορά σε σχέση με τους άντρε. και επίσης 40% διαφορά στη συντάξη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενώ η σύνταξη που είναι το αποκορύφωμα μιας μακράς εργασιακής ε, περίοδου και η μεγάλη συνταξιοδοτική διαφορά δείχνει ακριβώς ε, τις τεράστιες ανισότητες και διακρίσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. έχω μια πολύ σημαντική πρόταση που μερικώς τουλάχιστον θα, βελτίωσε, θα βελτίωνε την κατάσταση είναι το πακέτο για την εξορρόπηση της ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή. Αναφερθήκατε σε αυτό το πακέτο και είπατε ότι βρίσκεται σε, στο Συμβούλιο ε, για συζήτηση. Πώς θα ε, αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που το Συμβούλιο κατέληξε συμφωνία και οφείλω να εκφράσω τη μεγάλη μου απογοήτευση για το περιεχόμενο αυτή τη. ε, ε θέση του Συμβουλίου, γιατί δέχτηκε μόνο δεκαήμερη άδεια μεταποδοχών γονική. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεμονωμένο δικαίωμα για γονική άδεια μεταποδοχών και εσείς ε, είπατε ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ευρωπαϊκό, θα πρέπει να επιληθεί σε εθνικό επίπεδο. Οπότε τίποτα δεν αλλάζει τελικά, γιατί μόνο έξι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν καταβάλουν ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ για γονική άδεια. Ποια είναι η θέση της Αυστρίας, ε, γιατί εσείς ασκείτε την Προεδρία στο Συμβούλιο, οπότε ε, έχετε ε, μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε αναφαδόν υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ενώ η θέση του Συμβούλιο απέχει παρασάγκαση από την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενστερνίστηκε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι πολύ, σημαντικό, ε, πολύ σημαντική ψηφοφορία για το θέμα αυτό και ελπίζω η σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δούμε μετά πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας με το Συμβούλιο. Επίσης, ε, σίγουρα η βιομηχανία 4.0 θα είναι κινητήριος δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς ε, η αδιαφορία, οι, οι παραλήψεις που υπάρχουν στην πρόσληψη, στην απασχόληση των γυναικών για τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντική, πολύ περισσότερη από άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλους τέσσερις ομιλητές στον κατάλογο, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την κυρία Ρέγκνερ. και τον κύριο Πυρίνσκι. Επειδή είναι παρόμοιες θα προσπάσω να απαντήσω από κοινού. Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης. Η προσθέμενη αξία είναι όταν βοηθά στην εφαρμογή των διασυνοριακών δικαιωμάτων. Και αν ε, δούμε απτά, απτές βελτιώσεις ε, σε εθνικό επίπεδο και για τους εργαζομένους ε, και για τους εργοδότες. Σίγουρα πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν πάρα πολλά και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες. Υπάρχουν άλλοι φορείς, υπάρχουν ε, δομές ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και εδώ κάποια διπλή αρχή, αλληλεπικάλυψη, όλα αυτά θα πρέπει να τα μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε δομές ε, που θα λειτουργούν πάρα πολύ καλά και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ε, και να παραμείνουν ε, οι καλές δομές που ισχύουν, διότι είναι λογικό να δημιουργούμε μόνο δομές όταν δεν υπάρχουν. Σίγουρα θα πρέπει και για τη διασυνορική εργασία να έχουμε πιο αναλυτικές διατάξεις. Θέλουμε να βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να υπάρχει προστέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχο λοιπόν των διαπραγματεύσεων είναι η ευρωπαϊκή αυτή αρχή απασχόληση να συνιστά ε, προστιθέμενη αξία. Και εκεί λοιπόν θα ε, κάνω ό,τι μπορώ. Ω δεύτερη Ένα άλλο ερώτημα τη κυρία Ρέγνερ για τη συμφιλίωση προσωπική από ζωή. Έχουμε ε, στόχους και προτεραιότητες στην οδηγία. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη δέσμη μέτρων ε, για τη συμφιλίωση προσωπικής επαγγελματικής ζωής, ισότητα ανδρών και γυναικών, ε, ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και μείωση μισθολογικού σταδηματικού χάσματος. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε ε, υπόψη μας και τις νέες ε, ευέλικτες μορφές εργασίας. Σίγουρα θέλουμε να υπόψη μας ε, την ανάγκη για αγωνική άδεια, την άδεια όχι μόνο μητρότητας αλλά και άδεια πατρότητας. Πράγματι υπάρχει αυτό το δεκαήμερο της μεταποδοχών άδεια πατρότητας και 1,5 μήνας μεταποδοχών αγωνικής άδειας συγγένει. Τώρα ε, υπάρχει υπάρχουν διατάξεις ε, ε, που αφορούν την αύξηση της γονικής άδειας ε, ή για τα γονείς που έχουν παιδιά ως ηλικία 8 ετών. Προβλέπονται άλλες διατάξεις. Η προσπάθειά μας είναι να λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, είναι εξελίξεις που έγιναν σε επίπεδο δεκαετιών. διότι ό,τι αφορά ε, τις αποδοχές ε, για την ε, γονική άδεια. Το πιο επίμαχο ζήτημα εδώ είναι από πότε αρχίζει να υπολογίζεται, από ποια ημέρα αρχίζει να υπολογίζεται αυτό το επίδομα και υπάρχει στο θέμα αυτό στο Συμβούλιο διαφωνία. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε ε, να καταλήξουμε σε ένα πιο ευέλικτο μοντέλο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος για να μπορεί να προβεί το κάθε κράτος μέλος σε μια ρεαλιστική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ελπίζω σε συνεργασία μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του μέρους διαλόγου να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα άλλο ερώτημα της κυρίας ε, Ρέγνερ ήταν το gold plating, ο κανονιστικός περιθωρισμό. Υπάρχει task force για την επικουρικότητα και χθε ε, κατατέθηκε έκθεση συγκεκριμένα Υπάρχουν αρκετές νομίζω ρήτρε ε, που μπορούν να, ε, αποτελέσουν ε, εγγύηση για την αποφύγη αυτού του υπερθεματισμού. Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις και την αποφύγη καταχρήσεων, εδώ έχουμε πολλές προδιαγραφές και κανόνες σε επίπεδο κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις για την αποφύγη του κοινωνικού dumping. Υπήρξε και συμφωνία για αλλαγή, για τροποποίηση της σχετικής οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων πρόσφατα ε, και νομίζω ότι έχουμε ενισχύσει πλέον ένα πολύ καλό εργαλείο ε, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού ντάμπινγκ και επίσης άλλα θέματα όπως είναι η πρόσβαση, οι πληροφορίες, η διαμεσολάβηση, ο έλεγχος ε, των κρατών μελών είναι πλέον κατοχυρωμένα με την επικαιροποιημένη οδηγία. Και βέβαια τα κράτη-μέλη θα δουν κατά πόσον, ε, ε, μάλλον θα δούμε κατά πόσον υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων από τα κράτη-μέλη. Η Αυστριακή Προεδρία ε, επίσης και στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης θα φροντίσει στην εντολή της να είναι όλα αυτά πάρα πολύ ξεκάθαρα. Σε σχέση με την ερώτηση του ε, βουλευτού, ε, σίγουρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να καταλήξει τη θέση του. Στο Συμβούλιο επίσης ε, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τα επιδόματα που είπατε, ε, είχαμε ένα θέμα με το επίδομα ανεργίας και δεν καταφέραμε στο Συμβούλιο να καταλήξουμε ε, σε συμφωνία. Σίγουρα ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση επί του περιεχομένου και στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων ε, θα πρέπει να συζητηθούν ε, τα ζητήματα ένα προς ένα. Και εδώ σας ε, διαβεβαιώ ότι θα έχω την προσέγγιση της ουδέτερης διαμεσολαβήτριας και δεν θα υποστηρίξω την αυστριακή εθνική θέση. Έρχομαι στην κυρία Αρενά. Η Αυστριακή Προεδρία προσπαθεί να καταλήξει σε μια ισορροπημένη συμβαστική πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Θέλουμε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Σίγουρα αυτή είναι μια προτεραιότητα, ε, είναι ένα σημαντικός στόχος ε, ε, και μιλάω πάντα για τη δεκαήμερη άδεια πατρότητας και την άδεια τη γονική. Ε, που έχει διάρκεια 1,5 μήν. Σίγουρα, όπως είπα, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες ε, στα κράτη-μέλη. Μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Για τον κύριο Κώσα, πράγματι έχουμε προχωρήσει σημαντικά ήδη από την Βουλγαρική Προεδρία. Δεν έχουμε όμως ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα. Ε, τον ε, τομέα, ε, ένα σημαντικό θέμα είναι το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Πάντω το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την, τα άτομα με αναπηρία, για την οικονομία. Θεωρούμε το θέμα περί προσβασιμότητα προτεραιότητα για την Αυστριακή Προεδρία και ελπίζουμε μπορέσουμε να το κλείσουμε στη διάρκεια τη Προεδρία μα. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, ένα πολύπλοκο φάκελο και υπάρχει μια απόσταση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για την προετοιμασία και να μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε τις ε, διαβουλεύσεις μας ε, από το φθινόπωρο. Ε, για τους κυρίους Κώσα και Σόμπορ και την κυρία ε, Κατσόφσκα, Ραντεύσκα, κάπως έτσι λυπούμε αν δεν μπορώ να προφέρω σωστά τα ονόματα. Ε, πρέπει να πω ότι ε, δεν θέλω να μιλήσω για την εθνική θέση ό,τι αφορά την αποσαρμογή, την τιμαριθμική και ο συνάδελφος Στράους που ήταν παρόν σε μια άλλη επιτροπή χθε είπε τα σχετικά και πρέπει να πω ότι είμαστε ε, και εμείς σύμφωνοι και έχει συμφωνηθεί και το θέμα της αναπροσαρμογής, αναπροσαρμογής και ε, στο πλαίσιο των ε, διαβουλεύσεων για το Brexit και για το επίδομα τέκνου και για τα οικογενειακά επιδόματα. Υπάρχουν τα συστήματα συμμετρικής προσαρμογής που ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την κυρία Κοσλόφσκα, Ραγεύιτς. Πράγματι υπάρχει μισθολογικό ε, χάσμα. Ε, θέλουμε ε, να προωθήσουμε την γυναική απασχόληση, να αυξηθούν τα ποσοστά και βέβαια να αυξηθούν και αμοιβέ για την ψηφιοποίηση απασχόληση 4.0 και βιομηχανία 4.0. Έχουμε, όπως σας είπα, μια διάσκεψη το Σεπτέμβριο και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα εκεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.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 τα πράγματα αλλάζουν, ζητούμε συγγνώμη. Ε, συνδυασμός λοιπόν ψηφιοποίησης και ε, μετανάστευσης. Τι ακριβώς σκέφτεστε γύρω από αυτό. Ε, δεν προβλέπετε κάποιο θέμα και λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ε, από του βήματος θα μπορούσα ενδεχομένως διμερός μαζί σας να το συζητήσω. Κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλώς ήρθατε, Υπουργέ, στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε για όλα αυτά που θέλει να κάνει η Προεδρία σας στον κοινωνικό τομέα. Φοβάμαι όμως πως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ετοιμάζεστε να κάνετε στη χώρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον νόμο που σχεδιάζεστε νεοθετήσετε για την 12ωρη ημερήσια εργασία στη χώρα σα. Είμαι βέβαιη πως γνωρίζετε ότι η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία απαγορεύει κάτι τέτοιο. Έχετε συμβουλευτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υιοθετήσετε αυτήν την αλλαγή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Σε απάντηση που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε γραπτή ερώτηση στηρίζει πως οποιοδήποτε αλλαγές στον τομέα της εργασίας στα κράτη-μέλη πρέπει να επακούν στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παραπέμπτει επίσης σε έρευνες για την υγεία και την ασφάλεια στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, οι οποίες εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εσείς έχετε κάνει τις κατάλληλες έρευνες για την επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων το μέτρο που προτίθεστε να υιοθετήσετε. Θα ήθελα να μας διαφωτίσετε παρακαλώ γιατί έχουμε μεγάλη αγωνία από την είδηση. Thank you, Mr. Schuster. Ευχαριστώ, κύριε Σούστερ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι έχετε ε, την πρόσταση περιλάβετε στο θεματολόγιο και με τη διοργάνωση μια διάσκεψη του θέμα αυτό, το θέμα της ψηφιοποίησης και των σχετικών ε, συνεπειών. Ε, φαίνεται ότι ε, χρειάζεται ε, ρύθμιση το ζήτημα αυτό από θετική πλευράς, αλλά η Επιτροπή προς το παρόν πρέπει να περιμένει. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις οποίες εσείς σχεδιάζετε ενώ Νομοθετικέ νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ε, ε, σίγουρα αυτές προέρχονται από την Κομισιόν σε πρώτη φάση, όμως εσείς μπορείτε να πάρετε πολιτική πρωτοβουλία και να δώσετε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλετε το αίτημα να αναλάβει πρωτοβουλία νομοθετική. Τι ετοιμάζετε εσείς. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε γιατί ε, έχουν και άλλους δύο συνάδελφους που θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ε, στην κυρία Κούνεβα ότι την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ερώτηση, αλλά είναι μια ερώτηση που αφορά τα εθνικά ζητήματα, την εθνική πολιτική. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν προβλέπει κάποια συγκεκριμένη, κάποιο συγκεκριμένο όριο. Ε, προβλέπει βέβαια 48 ώρες ε, την εβδομάδα ε, για την ε, εβδομαδιαία ε, διάρκεια της εργασίας, αλλά μπορεί αυτή να αυξηθεί μέχρι τις 60 ώρες και μέσα σε τέσσερις μήνες 48. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, αλλαγές που έχουμε κάνει στην νομοθεσία μας ε, που δεν έρχονται σε αντίθεση, πιστεύουμε αυτές οι συγκεκριμένες που είπα, δεν έρχονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και όπως είπατε και εσείς κύριε Σούστερ για την νομοθετική πρωτοβουλία αυτή εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τις ε, συστάσεις μας ε, φυσικά θα μπορούσαμε να απευθύνουμε κάποια αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα και επίσης και το ζήτημα των νέων μελετών. Ότι χρειάζεται να είμαστε πιο ευέλικτοι ε, στην αγορά εργασία. Ε, αλλά υπάρχει το θέμα συμφιλίωση ε, τη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Θα το ψηφίσουμε εμεί στην Επιτροπή. Εσεί τοποθετηθήκατε από αυτού. Αναφέρατε και τη συγκεκριμένη οδηγία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα. Η συμφιλίωση προσωπικής επαγγελματικής ζωής είναι κάτι κεντρικό. Δεν θα έχει κάποιος ε, ο οποίος θα χρειαστεί στο μέλλον να εργάζεται 12 ώρες τη μέρα πολύ λιγότερο προσωπικό χρόνο. Δεν πρέπει να ληφθεί από αυτό υπόψη. Επίσης, ό,τι αφορά το ψηφιακό ε, τομέα αν αυξηθεί ε, το ωράριο εργασίας από τις 8 ώρες ε, σε πολύ περισσότερες, ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το πόσο υψηλή εξειδίκευση χρειάζεται στον τομέα αυτό της ψηφιοποίησης. Νομίζω ότι και ο κύριος Μπέκερ θέλει να κάνει μια τελευταία ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά επιδόματα. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Όλοι όμως ε, μπορούν να συνεισφέρουν. Ε, πρέπει να δώσετε, να ε, ενημερώσετε σωστά ε, για, το θέμα αυτό των οικογενειακών επιδομάτων. Τα οικογενειακά επιδόματα δεν ε, εντάσσεται στις κοινωνικές εισφορές. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ο εργοδότης ε, προκαταβολικά να καταβάλει α, ε, ως επίδομα ε, ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Και αυτό είναι ε, φυσιολογικό ότι πρέπει να έρθει να προσθεθεί στο επίδομα για το κόστος ζωής. Είναι όσο πιο υψηλό το, το επίδομα, τόσο λιγότερο πρέπει να είναι το πρόσθετο αυτό ποσό που πρέπει να δοθεί εξού και υπάρχει αυτό το ζήτημα της τιμαρτινικής αναπροσαρμογής που έχει προταθεί, έχει προταθεί και, για, και από τη Βρετανία. Ε, και το θέμα είναι τι θα γίνει με το, μετά τον Brexit. Ε, υπάρχει αυτή ε, η, πρόταση για την, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ε, αυτή η αρχή ε, θέλουμε να είναι στο δυνατόν πιο αποτελεσματική. Ποια είναι η άποψή σας ότι αφορά αυτούς τους ελέγχους στα κρατη Θέλετε να έχει η αρχή αυτή έναν ελεγκτικό ρόλο. Πόσο θεωρείτε ότι αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ απαντήσεις. Ε, για τον κύριο Τέτσιεν, για την ε, πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, τα έχω πει και είπα ότι είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές αυτά τα οποία προτείνουμε, γι' αυτό μην ανησυχείτε. Επίσης, ε, πρέπει να σας πω ότι, κύριε Μπέκερ, έχω έρθει σε επαφή και με την αρμόδια επίτροπο Τάισεν για το θέμα αυτό. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουν τεθεί οι ερωτήσεις μας, πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις. Θα είμαστε όσο πιο δραστήριοι μπορούμε κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. θα θέτουμε ερωτηματικά, αλλά θα θέλαμε να μας δίδετε και απαντήσεις. Από ό,τι φαίνεται από τη συζήτηση μέχρι τώρα ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα επανέλθετε ίσως και στην Επιτροπή μας, ενδιαφέρεστε για τις απόψεις μας ανάλογα με τα θέματα και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα. Πάντως ελπίζουμε ότι θα είστε μαζί μας και θέλω να ευχαριστήσω και τη διερμηνία που μας βοηθούν στην επικοινωνία. Αν και γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα και κάποια από σας απεργείται. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Thank